So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Επόμενο θέμα στη μέση διάταξη είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γιάννη Ρίχτερ, Υπουργό Εργασία Κοινωνικών Υποθέσεων και οικογένεια της Σλοβακίας. Κύριε Υπουργέ, καλωσορίσατε θερμά Εγκάρδια στην Ομιγυρίδα. Νομίζω για πρώτη φορά έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάσσουμε απόψεις με τη Σλοβακική Προεδρία στην Επιτροπή μας. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή. Η καιρή είναι δύσκολη αλλά και συναρπαστική ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά την απασχόληση και την εργασία, τις κοινωνικές υποθέσεις και λοιπά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε σημαντικές ε, υποχρεώσεις ενώπιόν μας που αφορούν και τη Σλοβακική Προεδρία. Μετά την εισαγωγική σας τοποθέτηση θα έχουμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε και σε συζήτηση χωρίς να μακρηγορώ και χωρίς μεγάλη εισαγωγή, Σας δίνω μέσα στο λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, θα ήθελα να σε ευχηθώ καλό απόγευμα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή για μένα το ότι βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, εκπροσωπώντας τη στοβαγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να αφαιρθώ στις βασικές προτεραιότητες τη Προεδρία όσον αφορά τους επόμενους μήνες. Η Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης της κοινωνικής πολιτικής, της πολιτικής απασχόλησης, των εργασιακών συνθήκων, καθώς επίσης και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς επίσης και της πολιτικής εκείνης που έχει να κάνει με την μετακίνηση και την κινητικότητα, των Ευρωπαίων εργαζομένων. Όλοι αυτοί οι διαφορετικοί κλάδοι έχουν να κάνουν με την ίδια τη ζωή προσωπική και επαγγελματική των Ευρωπαίων πολιτών. Είτε λοιπόν αναφερόμαστε για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, είτε μιλάμε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες απασχόλησης από συγκεκριμένου οργανισμούς, είτε μιλάμε για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, είτε μιλάμε για μετανάστες εργαζόμενους ή συνταξιδοτικά κοινωνικά δικαιώματα, όλα αυτά τα ζητήματα μας αφορούν άμεσα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πιστεύω ότι ε, οι κοινωνικοί εταίροι, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλές ομάδες συμφερόντων, αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις, δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα αυτά. Για παράδειγμα, τα συνταξιδοτικά δικαιώματα μας επηρεάζουν όλους, μας αφορούν όλους. Προσβλέπω λοιπόν σε μια επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας και πιστεύω ότι μέσω της συνεργασίας αυτής, μέσω των συνεχών επαφών που μπορούμε να έχουμε, μέσω της ανταλλαγής απόψεων, μπορούμε πραγματικά να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και την ποιότητα απασχόλησης των εργαζομένων και των Ευρωπαίων πολιτών, πράγμα το οποίο αποτελεί στόχο για όλους μας. Βασική προτεραιότητα στα, στον τομέα τη απασχόληση και τη κοινωνική πολιτική είναι η διασφάλιση των θέσεων απασχόληση, καθώ επίση και τη ευημερία για το παρόν και για το μέλλον. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η βασική προτεραιότητα πολλών τεχνικών και πολιτικών συνεδριάσεων που θα λάβουν χώρα και που θα ακολουθηθούν και από μία σειρά εκδηλώσεων στην Σλοβακία κατά τη διάρκεια βέβαια της Προεδρίας μας. Θα θέλαμε να επικεντρωθούμε κυρίως στην πρόθεση της αξιοπρεπούς εργασίας, στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και θέλουμε επίσης να επικεντρωθούμε και σε μέτρα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το άτυπο συμβούλιο ΕΠΣΚΟ, το οποίο θα λάβει χώρα, που έλαβε χώρα μάλλον στις 14 και 15 Ιουλίου στην Πρατισλάβα, ήταν η αρχική εκδήλωση για την Σλοβακική Προεδρία όσον αφορά τις προτεραιότητές μας στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων επικεντρωθήκαμε στις υφιστάμενες προκλήσεις, κυρίως όσον αφορά τις τεχνολογικές αλλαγές που επηρεάζουν βέβαια, που επηρεάζονται από τη μετανάστευση, από την γύραση του πληθυσμού, από τις δημογραφικές αλλαγές, από την ψηφιοποίηση και τις επιπτώσεις που όλα αυτά μπορούν να έχουν στην αγορά εργασίας. Οι Υπουργοί λοιπόν συμφώνησαν τότε ότι η ψηφιοποίηση και η ρομποτική επηρεάζουν πολύ σημαντικά την αγορά απασχόλησης. Ακριβώ επειδή έχουμε πάρα πολλέ τεχνολογικέ αλλαγέ, έχουν χαθεί πολλέ θέσει απασχόληση. Πολλοί άνθρωποι έχουν αντικατασταθεί από τι μηχανέ, από τα ρομπότ. Αλλάζουν επίση και οι απαιτήσει όσον αφορά τι δεξιότητε που θα πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι σε διάφορου τομεί. Ο ψηφιακό λοιπόν μετασχηματισμό τη οικονομία αλλάζει πραγματικά την ίδια τη φύση τη απασχόληση. Οι νέε μέθοδοι απασχόλησης απαιτούν και νέε δεξιότητες από τους εργαζόμενους. Η ψηφιοποίηση λοιπόν επηρεάζει άμεσα και την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Οι επιπτώσεις λοιπόν της ψηφιοποίησης στην αγορά εργασίας μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα κρίσιμες στο μέλλον στο πλαίσιο της κοινωνικής Ευρώπης. Εγκρίνοντα λοιπόν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τη σωστή πολιτική και λαμβάνοντα τις σωστέ αποφάσεις, νομίζω ότι είναι δυνατό να συμφιλιώσουμε την τεχνολογική πρόοδο με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των συζητήσεων που είχαμε, έγινε σαφέ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η ψηφιοποίηση να μην απευθύνεται μόνο στις τεχνικές πτυχές της απασχόλησης, αλλά θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και από το πρίσμα των κοινωνικών πτυχών της απασχόλησης προκειμένου να καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε στο επακρόν όλο το δυναμικό απασχόλησης που υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να έχω επ' αυτού και τη δική σας την συμμετοχή, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια κύριε Πρόεδρε και τη δική σας την Επιτροπή αλλά και τον ίδιο τον Πρόεδρο, εσάς κύριε Χέντελ, γιατί συμμετείχατε άμεσα στην άτυπη αυτή συνεδρίαση ΕΠΣΚΟ Πελεβεχώρα στην Πρατισλάβα τον Ιούλιο. Η Σλοβακική τώρα Προεδρία θα συνεχίσει τις εργασίες και τις διαπραγματεύσεις τη όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες εξετάζονται αυτή τη στιγμή σε τεχνικό, και, τεχνικό επίπεδο και επίπεδο εμπειρογνωμόνων στο Συμβούλιο. Θα κάνουμε κάθε τι το δυνατό προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο σε όλες αυτές τις νομοθετικές προτάσεις και να καταλήξουμε γρήγορα σε μία πολιτική απόφαση. Μία από τις πιο ευαίσθητες από πολιτικής πλευράς προτάσεις είναι η πρόταση για την απόσπαση των εργαζομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλύσει πλέον τις αντιδράσεις των 11 κρατών μελών που υπέβαλαν προτάσεις συγκεκριμένα τι προτάσει των 11 Εθνικών Κοινοβουλίων και αποφάσισε τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην τροποποιήσει την πρότασή τη. Η Σλοβακική λοιπόν Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επεξεργαστεί περισσότερο την πρόταση αυτή, θα έρθει σε επαφή με όλα τα κράτη-μέλη και στο πλαίσιο μια επικοδομητική συνεργασία θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική πρόταση. Το κείμενο λοιπόν της οδηγίας θα πρέπει να χαίρει υποστήριξης από όλα τα κράτη-μέλη. Η ομάδα εργασία του Συμβουλίου, η αρμόδια ομάδα εργασία, θα συνεχίσει τι εργασίε τη για το ζήτημα αυτό και θα ξεκινήσει την εργασία της ήδη από τις 2 Σεπτεμβρίου. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα είναι η τροποποίηση της οδηγίας όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων απέναντι στους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε, καρκίνογόνου και μεταλλεξιογόνου παράγοντες. Έχουμε έναν κατάλογο ουσιών που αναφέρονται πλέον στην πρόταση αυτή και που αποδεδειγμένα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Το να θέσουμε λοιπόν ανώτατα όρια για τις ουσίε αυτές και να τηρήσουμε τα όρια αυτά θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τον κίνδυνο έκθεσης των εργαζομένων σε αυτές τις ουσίες και παράλληλα θα συμβάλλει σε μια καλύτερη προστασία των εργαζομένων αυτών. Θέλουμε να συνεχίσουμε την πολύ καλή εργασία που έκανε για το ζήτημα αυτό η Ολλανδική Προεδρία και θα προσπαθήσουμε το στομότερο δυνατό να πετύχουμε γενική προσέγγιση σε επίπεδο Συμβουλίου και συγκεκριμένα στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ του Οκτωβρίου. Θα ενημερώσουμε ανοιχτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συνεργαστούμε με, τον αρμόδιο, με την αρμόδια μάλλον εισηγήτρια, την αντιπρόεδρο της Επιτροπής σας, την κυρία Μαρίτα Ουλτσκόκα, να καταφέρουμε να καταλήξουμε μαζί σας το στομότερο δυνατό σε μια κοινή συμφωνία. Θα ήθελα παράλληλα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την σταδιακή επικαιροποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, της, του συνόλου της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα υποβάλει μια πρόταση οδηγίας όσον αφορά τον δεύτερο κατάλογο καρκινοκόνων παραγόντων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Το ζήτημα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία θα μας απασχολήσει και στην τεχνική συνδιάσκεψη που θα λάβει η χώρα στις 24 και 25 Οκτωβρίου στην Πρατισλάβα. Και η οποία θα ασχοληθεί με την βελτίωση της πρόληψης στα πλαίσια μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας. Στόχος της συνδιάσκεψης αυτής είναι να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τους πολίτες όσον αφορά το ζήτημα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο απασχόλησης, καθώς επίσης και να αφαιρθούμε στις νέες δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να αποκριθούμε στις νέες τεχνολογίες και στις νέες μορφές απασχόλησης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη μας την γύρανση του ενεργού πληθυσμού. Μια άλλη σημαντική νομοθετική πρόταση στα πλαίσια της Προεδρίας μας είναι η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα. Από νομικής πλευράς πρόκειται για μια πολύπλοκη πρόταση. Στόχος της πάντως να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να καταρρύψει τα εμπόδια τα οποία εφίστανται αυτή τη στιγμή στο συνεργειακό εμπόριο και κυρίως να βελτιώσει την κατάσταση των ατόμων που έχουν αναπηρίες προωθώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες φιλοδοξία της Σλοβακικής Προεδρίας εν προκειμένου είναι να βελτιώσει και να τροποποιήσει το κείμενο αυτό προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και προκειμένου να μειωθεί τόσο το διοικητικό όσο και το χρηματοοικονομικό άκθος το οποίο βαρύνει τόσο τους επιθεωρητές όσο και τους οικονομικούς φορείς. Θα ασχοληθούμε όμως και με μη νομοθετικά ζητήματα. Και κυρίως αυτό που θα μας απασχολήσει είναι όλα αυτά τα ζητήματα που άπτονται των νέων. Ήδη από τον Οκτώβριο περιμένουμε μία έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει ως στόχο να αξιολογήσει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την εγγύηση των νέων και πώς έχει προωθήσει αυτό την απασχόληση των νέων. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την πρωτοβουλία αυτή και μετά το 2016. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ε, υψηλά ποσοστά ανεργία των νέων, να καταφέρουν να υποφεληθούν από την πρωτοβουλία αυτή. Η Σλοβακία βλέπει με πολύ θετικό πνεύμα την πρωτοβουλία αυτή, καθότι βασίζεται σε μια πολύ θετική εφαρμογή του προγράμματο αυτού σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό βοήθησε πραγματικά την ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας. Η Σλοβακική Προεδρία λοιπόν προτίθεται να επεξεργαστεί συμπεράσματα του Συμβουλίου προκειμένου να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τις συστάσεις αυτές και σε εθνικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό όμως να δούμε πώς θα καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε την πρωτοβουλία αυτή και μετά το 2016. Το ζήτημα της ε, ανεργίας των νέων και των ε, προοπτικών απασχόλησης των νέων θα μας απασχολήσει και σε μια συνδιάσκεψη που θα λάβει η χώρα στις 10 και 11 Οκτωβρίου του 2016, όπου θα επικεντρωθούμε στη βελτίωση της κατάστασης των νέων Ρωμά ως κινητήρια δύναμη αλλαγής. θα συμμετέχουν πολιτικοί βέβαια στη συνδιάσκεψη αυτή, αλλά το πιο σημαντικό είναι θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των ίδιων των Ρωμά, οι οποίοι θα είναι σε θέση να μας πούνε πώς έχουν τα πράγματα και πώς αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τις προκλήσεις της ε, μειονότητας των Ρωμά στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προβάλλουμε περισσότερο τις δραστηριότητες των νέων Ρωμά και θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Ρωμά σε ευρωπαϊκό, εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο. Το ζήτημα της ενσωμάτωσης των Ρωμά θα μας απασχολήσει και στα πλαίσια όμως του Συμβουλίου και θα θελήσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα του Συμβουλίου αυτή, αυτή τη στιγμή υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξη για του Ρωμά. Οι Ρωμά μολονότι αποτελούν μειονότητα, σίγουρα αποτελούν μειονεκτούσα ομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά ξεχνάμε πολύ συχνά ότι είναι πλήρει πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν τέτοια δικαιώματα και τι ίδιε υποχρεώσει με του υπόλοιπου Ευρωπαίου πολίτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε την κατάλληλη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να μην περιθωριοποιούνται οι Ρωμά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε τους ίδιους του Ρωμά στην επίτευξη λύσεων για τα προβλήματά τους. Ένα άλλο ζήτημα που πλήττει τις κοινότητες των Ρωμά είναι η μακροπρόθεσμη ενεργεία. Το ζήτημα βέβαια αυτό δεν απασχολεί μόνο τη μειονότητα των Ρωμά, θα έλεγα ότι είναι ένα οριζόντιο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττει πολλέ ομάδε στι κοινωνίε μα και βέβαια και τη Σλοβακία, η οποία αντιμετωπίζει το πρόβλημα τη μακροπρόθεσμη ανεργία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα συζητήσουμε το ζήτημα αυτό στα πλαίσια μια άτυπη συνεδρίαση Επιτροπή Απασχόληση, στα πλαίσια τη οποία θα θελήσουμε να θέσουμε τελικά ένα άτυπο πλαίσιο για την καλύτερη ενσωμάτωση των μακροπρόθεσμα ανέργων στην αγορά εργασία. Θέλουμε επίση να προωθήσουμε μια σειρά συζητήσεων μετά από συστάσει του Συμβουλίου και νομίζω ότι αυτό θα γίνει σε μια συνεδρίαση του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ στο Λουξεμβούργο. Θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια των Υπουργών Απασχόληση να δούμε πώ μπορούμε να μειώσουμε τα ποσοστά μακροπρόθεσμη ανεργία και πώ μπορούμε να προωθήσουμε την καλύτερη ενσωμάτωση των μακροπρόθεσμων ανέργων στην αγορά απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή λοιπόν η ανταλλαγή εμπειριών και πρωτοβουλειών μπορεί πραγματικά να εμπνεύσει και άλλα κράτη-μέλη προκειμένου να υιοθετήσουν θετικές πρακτικές. Προκειμένου να αυξήσουμε τα ποσοστά απασχόλησης, ιδίως ανάμεσα στις γυναίκες, θα πρέπει να προωθήσουμε και μια πολιτική εξισορρόπησης, συμφιλίωσης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Επ' αυτού θα πρέπει να έχουμε κατά νου τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, όπως γνωρίζετε, έχει υποβάλει μια σχετική πρωτοβουλία που έχει να κάνει με την εξορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Θα ήθελα λοιπόν να χαιρετήσω τις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για το ζήτημα αυτό της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αλλά και γενικότερα για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Ξέρω ότι η δική σας η Επιτροπή έχει υποβάλει μια πολύ σημαντική έκθεση και θεωρώ ότι θα καταφέρουμε με την πρόταση αυτή αλλά και με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώσουμε την κατάσταση των γυναικών και την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό επίση το νομικό και το πολιτικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιωθεί προκειμένου να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι πολύ συχνά οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες επιβαρύνονται με την φροντίδα όχι μόνο των παιδιών αλλά και άλλων εξαρτωμένων μελών. Η Σλοβακική λοιπόν Προεδρία θα διοργανώσει μία συνδιάσκεψη με τον εξή τίτλο «Συμφιλίωση, εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία». Η συνδιάσκεψη αυτή θα λάβει χώρα στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου στην Πρατισλάβα. Εμπειρογνώμονες θα συμμετάσχουν στη συνδιάσκεψη αυτή και θα συζητήσουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα εξυγχρονισμού της εφιστάμενης νομοθεσίας προκειμένου να έχουμε νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκριθούμε στις συναδειόμενες τάσεις που έχουμε στην αγορά απασχόλησης. Και άλλες όμως συνεδριάσεις θα γίνουν στην ε, Σλοβακία, επίσημες ή άτυπες, οι οποίες θα έχουν ως στόχο όχι μόνο να σημειώσουμε πρόοδο σε συγκεκριμένους χώρους πολιτικής, αλλά να καταφέρουμε γενικά να προβάλλουμε μια θετική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ευρωπαίους πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε και να προβάλλουμε τα απτά ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα πρέπει στη συνέχεια να εξηγήσουμε με τρόπο απόλυτα κατανοητό και σαφή προς Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία. Πολύ συχνά, δυστυχώς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προχωρούν σε μια στρέβλωση της κατάστασης ή δίνουν πολλές φορές μια παραπλανητική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ευρωπαίους πολίτες. Προβάλλουν μια παραποιημένη εικόνα για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργούν κατά αυτόν τον τρόπο ένα ιδιαίτερα αρνητικό πνεύμα στα πλαίσια των Ευρωπαίων πολιτών. Θεωρώ λοιπόν ως Υπουργό Απασχόλησης της Σλοβακικής Προεδρίας ότι μπορούμε μέσω των κοινωνικών υποθέσεων και μέσω των υποθέσεων που της απασχόλησης να προωθήσουμε μια θετική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ζητήματα που της απασχόλησης, που της κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να πραγματικά να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να δείξουμε προς Ευρωπαίους πολίτες ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτούς και ότι πρέπει να προωθηθεί ακόμα περισσότερο. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ για την εισαγωγή αυτή. Η διαδικασία στην Επιτροπή μας παγίως έχει ως εξή. Δίνουμε πρώτα το λόγο στους συντονιστές των διαφόρων πολιτικών ομάδων και στη συνέχεια σε ένα δεύτερο γύρο ε, μιλούν ε, τα υπόλοιπα μέλη μας. Κάνω ερωτήσεις και τοποθετήσει. Ο Ντέιβιτ Κάσα, πρώτος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Υπουργέ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και ήρθατε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής μας. Αναφερθήκατε στη μέτρα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Σλοβαγική Προεδρία καλείται να αξιολογήσει το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο για να προωθήσει την απασχόληση των νέων. Και για το δικό μου κόμμα, αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων προτεραιότητα. Είχαμε την οικονομική κρίση και αυτό το ένιωσαν και στο πετσί τους, όπου η ανεργία των νέων σοβεί περισσότερο σε κάποιες περιφέρειες και λιγότερο. Αλλού στη χώρα σας, ας πούμε, την ίδια τη Σλοβακία, Υπουργέ, αν δεν απατώμε, η ανεργία των νέων κυμαίνεται γύρω στο 25%. Με περιφερειακές διαφορές μπορεί να φτάσει και 40%. the... ε, ποια είναι η άποψη του Υπουργού, πώς μπορείτε να βρείτε αποτελεσματικούς τρόπους για να αντιμετωπίσετε την ανεργία των νέων, ιδιαίτερα σε περιφέρειες που είναι σαφές ότι μέχρι σήμερα πολιτικές ήταν Μάλλον ατελές φορές. Ευχαριστώ. Οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, η Γιώτα Στάιρουκ. Ευχαριστώ, Υπουργέ, που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας. Ακούσαμε από την τοποθέτησή σας ότι ασχολείστε σε μεγάλο βαθμό και με θέματα που μας απασχολούν μας στην Επιτροπή μας απασχόληση. Θα περίμενα να ακούσω πιο συγκεκριμένα μέτρα όμως Πώς το φαντάζεστε αυτό το θέμα της καταπολέμησης ενεργείας των νέων. Πειράματα έχουν γίνει πολλά ήδη. Με σχετική επιτυχία και με σχετική αποτυχία. Εσείς σε αυτά τι θέλετε να αλλάξετε και να βελτιώσετε. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την μακροχρόνια ενέργεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει μια ανακοίνωση σχετικά, τι προτίθεται συγκεκριμένα να ε, αναλάβει ως πρωτοβουλία η Σλοβακική Προεδρία, γιατί η μακροχρόνια ενεργεία είναι χρόνιο πρόβλημα σε ε, όλα τα κράτη-μέλη. Χαίρομαι που αναφέρεστε στις τεχνικές προόδους, τεχνολογικές και το πλαίσιο, τι γίνεται η ψηφιοποίηση στο μέλλον και πώς θα να ρυθμίσετε ε, την επιρροή τη στην αγορά εργασίας και τις επιπτώσεις που θα έχει στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών. Αυτά τα θέματα είναι εξίσου σημαντικά για μας, όπως και η δίκαιη κινητικότητα στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Ξέρω ότι δίστανται οι απόψει εδώ, αλλά σε τελική ανάλυση αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να είναι στο κέντρο ο άνθρωπος πάντα, ο εργαζόμενος και εργαζόμενοι, γιατί ορισμένοι ε, είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης ε, στις ε, χώρες. Η απόσπαση εργαζομένων είναι ένα παράδειγμα και μόνο, υπάρχουν και άλλα. Στερούνται δηλαδή και τα βασικότερα εργασιακά τους δικαιώματα. Εκεί θα πρέπει να δουλέψουμε. Να μην έχουμε κούρσα ανταγωνισμό προς τα κάτω για το φθηνότερο εργατικό δυναμικό, αλλά για τις καλύτερες θέσεις εργασίας, τις πιο ποιοτικέ. Και έτσι βοηθούμε όλα τα κράτη-μέλη και δεν μπαίνουμε σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ μας. Χαίρομαι που θέλετε να εργαστείτε ε, για μια θετική Ευρώπη, μια αισιόδοξη Ευρώπη που να μην έχει ε, στο μυαλό της μόνο την ανθούσα οικονομία και τη συγκυρία σε όλα τα κράτη-μέλη Σημαντικά είναι αυτά, αλλά εξίσου σημαντικοί είναι και οι άνθρωποι που ζουν στην Ευρώπη. Όταν μας λέτε ότι ε, δημιουργούν κακή εικόνα τα μέσα ενημέρωσης και διαδίδουν τέτοια πράγματα, μήπως φταίνε καμιά φορά και οι πολιτικοί, άντρες και γυναίκες, των οποίων οι δηλώσεις απλώς μεταφέρονται από τα μέσα ενημέρωσης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και στο δικό μας πρόσωπο έχετε έναν έντιμο εταίρο για την ε, προσπάθειά σας στην κατεύθυνση αυτή. Η κυρία Τρεμπέσιους από το ΙΣΙΑ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την ε, εκτενέστερη παρουσίαση της ε, Σλοβακικής Προεδρίας. Αναφερθήκατε σε πολλά θέματα και εγώ θα ήθελα να σταθώ στα θέματα που απασχολούν την Επιτροπή μας, την Επιτροπή Απασχόλησης, την ανεργία δηλαδή των νέων, τους ε, μακροχρόνια άνεργους κτλ. Πιστεύω πως συμφωνούμε ότι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης είναι ιδιαίτερα σημαντική και είναι ταυτόχρονα μια μεγάλη πρόκληση στα πλαίσια της Προεδρίας της Σλοβακίας, εσείς πού βρίσκετε ότι υπάρχει ε, περιθώριο, πολιτικό περιθώριο για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις στήριξης της καινοτομίας που θα δημιουργήσει με τη σειρά της ε, θέσης απασχόλησης και εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς μπορούμε να γίνουμε προορατικοί. Για παράδειγμα, πώς μπορούμε να παραμερίσουμε τα εμπόδια που ε, στέκονται στον δρόμο της ε, ανάπτυξης θέσεων απασχόλησης. Επίσης, κάτι που θεωρώ εξίσου σημαντικό, υπάρχει μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βελτίωση των συνθήκων για τα άτομα με αναπηρία. Για παράδειγμα, η δημιουργία συγκεκριμένων υπηρεσιών η ευκολία στην πρόσβαση των ε, ανθρώπων αυτών σε συγκεκριμένα προϊόντα. Πιστεύουμε πως θα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Μπορούν να είναι ενεργοί επαγγελματικά και κοινωνικά. Υπάρχει κάποιο σχέδιο, μπορείτε να μου πείτε κάποια πράγματα περισσότερο για αυτό το θέμα, διότι αναφερθήκατε επιγραμματικά ποια εμπόδια βρίσκετε εσείς και πώς μπορούμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξουμε τις προσπάθειές σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Μάριαν Χάρκιν για την ομάδα Άλντε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ στην Επιτροπή μας. Θα χαρώ για τη μελλοντική μας καλή συνεργασία. Παρατηρώ το γενικό πρόγραμμα και διακρίνω τρία διαφορετικά στοιχεία. Αποτελέσματα, αποφυγή του κατακαιρματισμού και εστίαση στους πολίτες. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην ανάγκη να δείξουμε στους πολίτες ότι τα κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν θετικά αποτελέσματα. Το είπατε και ο ίδιος και πιστεύω πως συμφωνούμε όλοι για το πόσο σημαντικό είναι αυτό, διότι πολλά από αυτά που κάνουμε δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά. Εσείς έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση για το πώς ε, σκοπεύετε να ενημερώσετε τους πολίτες για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα, Όσον αφορά τις δεξιότητες και την απόσπαση εργαζομένων, η Μαρτίνα θα αναφερθεί σχετικά. Έχω όμως κάποιες άλλες ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στην πράξη για την προσβασιμότητα και την επιθυμία σας να προχωρήσει. Αναφερθήκατε στην τροποποίηση του κειμένου έτσι ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και να μειωθεί ε, ο διοικητικός εφόρτος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θεωρώ πως η πράξη για την προσβασιμότητα αφορά περισσότερο την απαλληφή των φραγμών για τα άτομα με αναπηρία, κάτι που όπως γνωρίζετε ε, είναι πακτό και οι αριθμοί τους αυξάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, αναφερθήκατε σε νομοθετικές αλλαγές στην εσωτερική αγορά, την, ε, τον συντονισμό των ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, την μετακίνηση των εργαζομένων. Υπάρχουν προτάσεις βέβαια, αλλά στα πλαίσια του Brexit έχουν αλλάξει πολλά. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι ισχύει τώρα, τι προτάσεις ε, υπάρχουν, ποιες προτάσεις δεν συζητιούνται πια, ποιες προτάσεις ε, αν υπάρχουν είναι καινούριε. Έπειτα, η εγγύηση για τους νέους, ε, υπάρχουν αποτελέσματα και τέλος, δεν αναφέρατε την συνεταιριστική οικονομία και ήλπιζα η Προεδρία της χώρας σας να συμπεριλάβει στο θεματολογιό της ε, την οικονομία αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Ρωνιακάρη για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ που μας αναφέρατε το πρόγραμμα της Προεδρίας της Σλοβακίας για τους επόμενους έξι μήνες. Και πιστεύω πως είναι αρκετά ωφέλιμος αυτός ο άμεσος διάλογος που έχουμε με το Συμβούλιο. Έχω μια ερώτηση σχετικά με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Αναφερθήκατε εν συντομία, όμως θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιες είναι οι θέσεις της Προεδρίας και ποιες οι προσδοκίες της στις ε, διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε βέβαια το αποτέλεσμα, όμως πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και τώρα μια γενικότερη ερώτηση για το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Επιτροπή μας τον Ιούνιο ψηφίσαμε μία έκθεση σχετικά με αυτό και τον Σεπτέμβρη θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Η έκθεση αυτή αφορά τις ε, συνθήκες εργασίας. Θέλουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Εσείς ε, τι σχέδια έχετε για την οδηγία, για την απόσπαση εργαζομένων, πώς μπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για τους πολίτες και τι συμβαίνει με τους ε, κοινωνικούς εταίρους, θα συμπεριληφθούν στις διαπραγματεύσεις ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η οχι ευχαριστω Λαμπερτό από τους Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να... Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό που ήρθε σήμερα και να ευχαριστήσω και την συνάδελφο Χάρκιν, η οποία αναφέρθηκε στο ότι υπάρχει ανάγκη να ενημερώσουμε τους πολίτες για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς ε, δεδομένων των ε, συνθήκων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα κάποια σχόλια από εσάς για το ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες ε, στον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Κάτι το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία διαβούλευσης. Τι συμβαίνει λοιπόν με την σχετική πρόταση. Με ενδιαφέρον επίσης άκουσα όσα είπατε για το σχέδιο για την κοινωνική συμπερίληψη των Ρωμά και για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Μάλιστα πίστευα πως αυτό ήταν κάτι που ήθελαν όλοι οι υπουργοί να αποφύγουν παρά να το προχωρήσουν. Υπάρχει η διάσταση πλέον της πρόληψης, η διάσταση για τις νέες δεξιότητες, για τη μετάβαση, την τεχνολογική μετάβαση σε μια ψηφιακή οικονομία. Στην Επιτροπή μας όμως εξετάζουμε αυτήν την μετάβαση από τη σκοπιά ε, της ε, επάρκειας των πόρων, της επάρκειας ενέργειας, το πώς δηλαδή θα αλλάξει η οικονομία και θα γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον, πιο αηφόρος. Θα ήθελα λοιπόν να κάνετε κάποια σχόλια για το πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτός ο τομέας, ε, πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι δεξιότητες, ποιες είναι οι νέες ανάγκες που θα προκύψουν στο τομέα αυτό. Να επαναλάβω και εγώ ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας και να προτείνουμε νέες ιδέες, διότι πιστεύω πως δεν δίδεται ιδέουσα προσοχή στο θέμα αυτό και εμείς ως Επιτροπή Απασχόλησης έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευτυχή. Δεν βλέπω την κυρία Τζέα, ούτε τον Ντομενίκ Μαχτά, οπότε πάμε ε, αμέσως στον επόμενο γύρο για να ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις. Η κυρία Μόρα Σάρτια, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ που μας κάνετε την τιμή να μας επισκέψετε εδώ στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσετε το πρόγραμμα της Σλοβακικής Προεδρίας. Τρεις ερωτήσεις έχω εγώ να σας κάνω. Πρώτη, αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Ξαναβρίσκεται μπροστά σας ένα πρόβλημα που είχατε εντοπίσει και στο παρελθόν, να αποφύγετε τους κατακαιρματισμούς. Τι θα κάνετε στο Συμβούλιο, με ποια μέθοδο θα το προωθήσετε, γιατί μέχρι τώρα ακούμε μάλλον για αντιστάσεις και αντιδράσεις με τη διαδικασία της κίτρινης κάρτας. Παρά για πραγματική βούληση να προωθηθεί αυτή η υπόθεση η οδηγία αυτή είναι από τα βασικά θεμέλια της κοινωνικής Ευρώπης. Το δεύτερο αφορά την εξέλιξη ε, την επαγγελματική. Τα δέκα επαγγέλματα που προσλαμβάνουν τους περισσότερους ε, εργαζομένους σήμερα δεν υπήρχαν πριν από δέκα χρόνια. Βλέπουμε ότι είναι λοιπόν ε, μία κούρσα ταχύτητας που πρέπει ε, να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Αλλιώς θα πρέπει κάθε φορά να τρέχουμε, να βρίσκουμε τα νέα επαγγέλματα και να μετεκπαιδεύουμε τους ανέργους μας. Και τι γίνεται επίσης με τα κοινωνικά ταμεία που βοηθούν στην επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Είστε διατεθειμένος ε, να ε, τα υπερασπιστείτε αυτά με νύχια και με δόντια έτσι ώστε να μην συνενωθούν και μην συγχωνευθούν με τα ταμεία συνοχής αλλά να μείνει ο άνθρωπος πραγματικά στο επίκεντρο όλης μας της προσπάθειας και της προσοχής. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω εδώ και που αναφερθήκατε σε όλα τα βασικά σημεία και τις προτεραιότητες της Προεδρίας. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, δεν μπορώ να αποφύγω να ρωτήσω για την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Είπατε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κάποια συνένεση. Στη σημερινή κατάσταση έχουμε από τη μια 11 κίτρινες κάρτες και από την άλλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εξακολουθεί να επιμένει στη δική της άποψη. Εσείς πώς θα το λύσετε αυτό, πώς θα το οδηγήσετε σε μια απεμπλοκή. Υπάρχει πρόταση για να προχωρήσουμε συνενετικά και πότε προτίθεστε να καταθέσετε τέτοια πρόταση για την εφαρμογή της οδηγίας του 2014, γιατί υπήρξε και καταληκτική ημερομηνία του 2016. Τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν με την οδηγία, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει καμία μελέτη αντικτύπου για το πώς εφαρμόζεται. Δηλαδή, να κάνουμε μία αποτίμηση πώς πήγε μέχρι τώρα η εφαρμογή πριν προχωρήσουμε στην επόμενη οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Και μια δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με την εναρμόνιση των επαγγελματικών, μάλλον την, να το πω αλλιώς, ε, τη συμφιλίωση ε, του επαγγελματικού με τον οικογενειακό βίο ή της επαγγελματικής ε, ζωής με το χώρο που έχει ο κάθε εργαζόμενος για ξεκούραση και αναψυχή. Ορισμένοι λέγουν ότι εμείς δεν αξιολογούμε αρκετά και δεν εκτιμούμε την εργασία των γονέων. Μπορεί ένας γονιός να δουλεύει, αλλά ένας γονιός που δεν δουλεύει και είναι σπίτι και αυτός δουλεύει. Και ε, συχνά δεν αξιολογούμε το ρόλο των γονέων στην ανατροφή των παιδιών, για παράδειγμα. Ε, σκέφτεστε να το λύσετε αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω, τη συμφιλίωση οικογενειακού με τον επαγγελματικό βίο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πλίνκεβιτσούτε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα στην Επιτροπή μας. Η Σλοβακία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια δύσκολη περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη σας Προεδρία. Ολόθρεμα λοιπόν σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Και ελπίζω ότι μαζί σας θα καταφέρουμε πραγματικά να ενισχύσουμε την κοινή μας ευρωπαϊκή οικογένεια. Καταβάλαμε πάρα πολλές προσπάθειες σε πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την απασχόληση των νέων. Έχουμε πλέον το πρόγραμμα για την εγγύηση των νέων, με ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο. Δεν πιστεύετε όμως κύριε Υπουργέ ότι υπάρχουν τελικά ακόμα πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι ακόμα δεν καταφέρουν να βρουν μια θέση απασχόληση και αναγκάζονται τελικά είτε να φύγουν από τη χώρα τους ή να εγκαταλείψουν ακόμα και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι ακόμα, δεν ασχολούμεθα και με το ζήτημα της ένδυας της φτώχειας των παιδιών. Ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν κάτω από το όρο της φτώχειας η κατάσταση είναι πραγματικά απέσια. Γίνεται κάτι από τη Στοβαική Προεδρία ή προτίθεται η Σλοβακική στοβαικη προεδρια να κάνει κάτι. Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο εν μέρει το κάλυψαν και αδελφή μου έχει να κάνει με το ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Επιτροπή Απασχόληση και η Επιτροπή για τη Δικαιώματα των Γυναικών έχουν υποβάλει μια κοινή πρόταση όσον αφορά την εξορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα διοργανώσετε μια συνδιάσκεψη το Σεπτέμβριο για το ζήτημα αυτό. Ωστόσο, τι πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε συγκεκριμένα χειροπιαστά κατά τη διάρκεια της δικής σας προεδρίας, προκειμένου να έχουμε μια ουσιαστική συμφίλιωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθυνθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας της να παρουσιάσει τέσσερα Σχέδιο οδηγιών, τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικά και ουσιαστικά για την εξορρόπηση επαγγελματική και προσωπική ζωή. Και η τελευταία μου ερώτηση, η δική μου χώρα, η Λιθουανία, ταλανίζεται αρκετά από την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Η Λιθουανία και όμορες τις χώρες έχουν μπλοκάρει αυτή τη στιγμή την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Δεν πιστεύετε πάντως εσείς ότι κατά τη διάρκεια της δικής σας προεδρίας θα πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες συζητήσεις για να καταλάβουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το μπλοκάρισμα τελικά, για ποιο λόγο τα κράτη-μέλη δεν συμμορφώνονται με την οδηγία αυτή ή γιατί τουλάχιστον δεν προβλέπουν ισότιμους μισθούς για κατηγορίες εργαζομένων όπως για παράδειγμα οι οδηγοί φορτηγών κατηγορίες επαγγελματικέ για τι οποίε θα πρέπει να προβλέπετε μια ισότιμη μισθολογική αντιμετώπιση. Χρειάζεται πρόεδρος για, για όλα αυτά τα σημεία. Γέριος, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, Υπουργέ. Εξ ονόματος, να και από μέρους μου, μάλλον, ε, σας έχω κάθε επιτυχία, εδώ κάθομαι, δεν με βλέπετε. Ε, η Ολλανδική ε, Προεδρία παρέδωσε σε εσά πλέον τη σκητάλη και μαζί με αυτή τη σκητάλη και κάποια προβλήματα που δεν κατάφερε να λύσει η ίδια. Χάρηκα όταν σας άκουσα να λέτε ε, ότι τα κοινωνικά θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την εικόνα που σχηματίζουν οι Ευρωπαίοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ απολύτως. Έτσι τα βλέπω και εγώ τα κοινωνικά ζητήματα. Οπότε νομίζω ότι είναι καλή αφετηρία αυτή. Έχω μια ερώτηση. Σας άκουσα να λέτε κάτι για τις 2 Σεπτεμβρίου. Ότι συνεδριάζει η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την απόσπαση των εργαζομένων, για την αντίστοιχη οδηγία. Έχετε καμιά ιδέα ή καμιά εικόνα για το τι θα συζητηθεί και τι θα διαμευθεί και είστε αισιόδοξο ότι θα μπορέσει να κλείσει το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της δικής σας προεδρίας. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει συνένεση και συμβιβασμή, αλλά σας ρωτάω πώς το βλέπετε εσείς, ποια είναι η δική σας εκτίμηση. Και κάτι άλλο που έχει σχέση με αυτό, κατά πολέμηση της την αναφέρετε, αλλά δεν αναφερθήκατε καθόλου σε κάποιες στρατηγικές που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε έτσι ώστε να ε, αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που έχουν σε πολλά μέρη εργαζόμενοι στην Ευρώπη ε, που έχουν πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη. Γιατί η ζωή είναι ακριβή και ε, ο κόσμος μπορεί να μην είναι άνεργος και παρόλα αυτά να είναι φτωχό και να μην μπορεί να ανταπεξέρχεται ε, στις ανάγκες του. Τι ε, σκέφτεστε να κάνετε εκεί ε, στα πλαίσια και του κοινωνικού διαλόγου για αύξηση των μισθών στην Ευρώπη, όχι μόνο κατά πολέμηση ενεργείας και της φτώχειας. Ευχαριστώ. Κούκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα και εγώ να σα καλωσορίσω στη σημερινή μα συνεδρίαση. Όπως είπε και ο Πρόεδρός μας στην αρχή της συνεδρίασής μας, εμείς, μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται για να συζητάμε θέματα απασχόλησης με τους υπουργού της κάθε Προεδρίας. Θίξατε διάφορα τέτοια ζητήματα κι εσείς ε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων η κυρία Σόροντοβα αναφέρθηκε στα προβλήματα τα οποία συναντούμε. Αν πραγματικά θέσουμε ως στόχο να καταφέρουμε να βρούμε μια συνετική πρόταση με την οποία να συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη, μάλλον αυτό θα είναι υπερφιλόδοξο. Ας θέσουμε καλύτερα πιο ρεαλιστικούς στόχους. Οι θέσει των κρατών μελών αυτή τη στιγμή διήστανται. Σας ρωτώ λοιπόν, η δική σας η Προεδρία έχει μια κάποια στρατηγική, τακτική, πώς να το θέσω ακόμα και κάποιο μυστικό όπλο ή συνταγή προκειμένου να καταλήξει σε μια συμβαστική θέση, μόνο και μόνο αυτό θα ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα. Δεύτερο ερώτημα. Η σλοφακικη Προεδρία αναφέρει ανάμεσα στις προτεραιότητές της και την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων. Ως προς αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι σχετικό πώς μπορείτε να βοηθήσετε και τους πιο ηλικιωμένους και κυρίως τους πιο ηλικιωμένους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη της λεγόμενης ε, αργυρής οικονομίας, αυτή δηλαδή που έχει να κάνει κυρίως με την τρίτη ηλικία. Πώς μπορούμε αυτή τη στιγμή να καταρρύψουμε κάθε μορφή διάκρισης που υπάρχει κατά των ηλικιωμένων εργαζομένων. Εύχομαι πραγματικά κάθε επιτυχία σε εργασία σας. Ευχαριστώ, κύριε Μαρτίνα Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Καλώς ορίστε στην Επιτροπή μας. Είμαι περήφανη που μπορώ αυτή τη στιγμή να συνομιλώ μαζί σας που προεδρεύετε του Συμβουλίου όσον αφορά την εγγύηση για τους νέους. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ζήτημα αυτό το θεωρείται προτεραιότητα τη Κυριακή Προεδρία, που είπε ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την πρόταση αυτή, το ότι πρέπει πραγματικά να δούμε ποιες ε, είναι, ποια είναι η πρόοδο που ενδεχομένω να έχει επιτευχθεί με το πρόγραμμα αυτό, αν είχαμε δηλαδή συγκεκριμένα αποτελέσματα, προτού αυξήσουμε τη χρηματοδότηση του προγράμματο. Αν δούμε τις ε, συστάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, που ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό, νομίζω ότι και αυτό θα συμβάλλει πολύ επικοδομητικά στην εργασία μας. Και υπάρχει και μία ακόμα διάσταση στο ζήτημα, οι δεξιότητες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε τις δεξιότητες και την απαιτούμενη γνώση να τις συνδέσουμε με τις απαιτήσεις της ίδιας της αγοράς εργασίας. Αυτή τη στιγμή έφτασα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ασχολούμαι με το ζήτημα αυτό εκτενέστατα και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα και τι επιχειρήσει. Νομίζω ότι οι εργοδότε θα πρέπει να συνεργάζονται περισσότερο με τι αρμόδιε εθνικέ αρχέ που καταρτίζουν τα προγράμματα εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων. Εσείς έχετε μια σχετική εμπειρία. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν θετικό να καταφέρουμε να εντατικοποιήσουμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στα κράτη-μέλη και να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών. Πώς μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις νέες δεξιότητες. Μπορείτε και από αυτού να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Και κάτι ακόμα, το κάλυψαν αυτό και άλλοι συνάδελφοι. Οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Κατά τη διάρκεια τη προηγούμενη Προεδρία, οι χώρε του Βίζεγκράτα είχαν πει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ε, ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Η Σλοβακία συγκεκριμένα έστειλε συγκεκριμένε συστάσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση τη οδηγία αυτή. Εμεί θεωρούμε ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει συζήτηση και θα ήθελα πραγματικά να, να γνωρίζω, όπως είπε και ο κύριος Κούκαν, αν έχετε κάποια μυστική συνταγή προκειμένου να καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο στα πλαίσια του Συμβουλίου. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες παρεμποδίζουν την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Κύριε Ριμπέρο, ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω στην ε, πρώτη μας συνάντηση και ελπίζω να ακολουθήσουν και πολλές άλλες. Ε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας. Έχω τις εξής δύο ερωτήσεις. Πρώτον, τι γίνεται με την εικόνα που έχουν οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει κάπως να διαφημίσουμε, την προβάλλουμε την Ευρώπη. Αυτό το καιρό εγώ είμαι εισηγήτρια του Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα της απασχόλησης και τα κοινωνικά. Το Κοινοβούλιο το Μάρτιο ήταν σαφέστατο στη θέση του και την άλλη εβδομάδα ε, θα έρθει και η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θέλουμε να υπάρχει μια ισορροπία στην Ευρώπη ανάμεσα ε, στην οικονομική και την κοινωνική διάσταση. Οι διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουν με διαφορετικό τρόπο. Και ο τρόπος ε, που βλέπουμε εμείς τα πράγματα, η αντίληψη που έχουμε εμείς για τα πράγματα είναι διαφορετική από εκείνη του Συμβουλίου. Όταν γυρνάμε στις χώρες μας, μας κατακλείζουν διάφορες ε, οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές, κανόνες, υποδείξεις, αλλά χάνεται κάπου εκεί η κοινωνική διάσταση. Θα πρέπει να βρεθεί ε, άλλος τρόπος συνεργασίας του ΕΠΣΚΟ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί οι πολίτες τι διαπιστώνουν. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λυσάει κυριολεκτικά για τα οικονομικά ζητήματα, αλλά αν χαθούν οι άνθρωποι και τα κοινωνικά ζητήματα, τι να τους κάνουμε τους αριθμούς και την οικονομία. Θα πρέπει να συνεχιστεί η κοινωνική προστασία και η ευημερία που έχουμε στην Ευρώπη Κοιτάξτε τι ψηλά ποσοστά ενεργείας αντιμετωπίζουμε, ιδιαίτερα για την ανεργία των νέων και για τη μακροχρόνια ανεργία. Ο πληθυσμός ε, γυράσκει, υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα, τα οποία δεν αφορούν μόνο τους νέους σήμερα ή τις μελλοντικέ γενιέ, αλλά και τις σημερινές. Άρα λοιπόν η κοινωνική Ευρώπη είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να διαφυλάξουμε και θέλω να σας ρωτήσω τι πρόκειται να κάνετε για να υπερασπιστείτε και να διατρανώνετε και την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχομαι τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό. Brexit. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσετε να προετοιμάζεστε για τις διαπραγματεύσεις με ε, τη Βρετανία. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους πολίτες των χωρών μας που εργάζονται σήμερα ε, στη Μεγάλη Βρετανία. Να προστατευθούν. και το αντίστροφο, Βρετανοί πολίτες που εργάζονται στις χώρες μας. Να γίνεται δημόσια συζήτηση, όχι σε κλειστά γραφεία και ιδιαίτερα γραφεία υπουργικά. Θέλετε να μα πείτε κάτι και για τον Brexit, τι στρατηγική έχετε. Ευχαριστώ. Θυμίζω το δίλεπτο που έχει ο καθένα στη διάθεσή του. Ο Άνταμ Κόσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Ακούσαμε επανειλημμένως το θέμα της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων και ότι δεν υπάρχει συνένεση αυτή τη στιγμή μεταξύ των κρατών μελών. Είναι ένα ζητούμενο. Και θέλω να σας ρωτήσω και εγώ για αυτό το θέμα. τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση και ένα δεύτερο τι γίνεται με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εργασία. Η Ολλανδική Προεδρία είχε κάποιες επιτυχίες. Θα τις συνεχίσετε εσείς. Ε, τι συγκεκριμένους στόχους έχετε και τι συγκεκριμένα σχέδια. Τι έχετε προγραμματίσει ως Προεδρία να κάνετε για το θέμα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία το επόμενο εξάμεινο. Και δεν αναφορά αποκλειστικά τους ανθρώπους με αναπηρία το θέμα της πρόσβασης σε προϊόντα και ε, υπηρεσίες είναι κάτι πολύ γενικότερο. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Μπενιφέ. Uh, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε για άλλη μια φορά δυνατότητα να σας ξανασυναντήσω. Σας συνάντησα μια πρώτη φορά στην Πρατισλάβα, uh, στα πλαίσια της επίσημης αντιπροσωπείας μας στην Πρατισλάβα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τον λόγο σας αυτό, για τις παρατηρήσεις που κάνατε. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο σε πάρα πολλά διαφορετικά ζητήματα. Θα ήθελα να σας ζητήσω την άποψή σας για την δυνατότητα, την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένα ταμείο επιδοτήσεων όσον αφορά τις χώρες εκείνες οι οποίες πλήττονται από ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας. Ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να λειτουργήσει στα πλαίσια οικονομικών κρίσεων για τις χώρες εκείνες που έχουν ένα κοινό νόμισμα και θα μπορούσε να ενισχύσει την εσωτερική ζήτηση και να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες ελληνικής. Ο Υπουργός Οικονομικών Παντοάν, ο Υπουργός Οικονομίας Ιταλίας, είχε κάνει μια σχετική πρόταση βασιζόμενο στις υφιστάμενες συνθήκες. Δεν ξέρω λοιπόν αν θεωρείτε ότι είναι σημαντικό από πολιτική και μακροοικονομική πλευρά σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Εγώ πιστεύω πω ναι, γιατί θα δείξει προ Ευρωπαίου πολίτε ότι λαμβάνει συγκεκριμένη δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση μια κοινωνική Ευρώπη. Η Σλοβακική λοιπόν Προεδρία προτίθεται να εμβαθύνει περισσότερο τι συζητήσει για αυτό το ζήτημα, θα συνεργαστεί περισσότερο με τι εθνικέ κυβερνήσει θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό και με παραμφερή ζητήματα, καθώς επίσης και με τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου ταμείου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, Χάβι Λόπε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, Υπουργέ. Χαιρόμαστε για την παρουσία σας εδώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι για την ψηφιοποίηση που αναφέρατε και εσείς στην αρχική σας τοποθέτηση και ποια είναι η συγκεκριμένη στρατηγική που έχουμε απέναντι σε αυτή τη διαδικασία που τη γνωρίζουμε πολύ καλά και μας απασχολεί εδώ. Και υπάρχουν μελέτες που τη χαρακτηρίζουν την ψηφιοποίηση και ως απειλή για την αγορά εργασίας. Κινδυνεύουν 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας από τη ρομποτική και μόνο ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ακούγεται. Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία ε, και για την παγκοσμιοποίηση και ε, για την, τις ελεύθερες συναλλαγές από την οποία επωφελούνται κάποιοι στην κοινωνία αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικά στρώματα και πολυπληθεί στην κοινωνία που πέφτουν θύματα και τελικά είναι χαμένοι και της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης. Και αυτό έχει επιπτώσεις και στην εκλογική συμπεριφορά του κόσμου από εκεί και πέρα. Λοιπόν, πώς σκεφτόμαστε να αντισταθμίσουμε τα αρνητικά. Δεν λέω, είναι, έχει και θετικά η ψηφιοποίηση, βεβαίως και θα τα αξιοποιήσουμε και θα τα εκμεταλλευτούμε, αλλά πώς θα υπάρχει μια στοιχειώδης ασφάλεια και αξιοπρέπεια για τους εργαζόμενους. Πώ θα γίνει αυτό με κοινωνικού μηχανισμού. Γι' αυτό μιλάμε εμεί εδώ για τον κοινωνικό πυλώνα. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί ξεκάθαρα, η Επιτροπή του κ. Γιούνκερ, η δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή εργάζεται από αυτού και θέλουμε να ακούσουμε συγκεκριμένε ιδέε για το τι θα κάνετε του επόμενου μήνε τη Προεδρία σα για να αναπτυχθούν αυτοί οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί σε ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό πλέον πυλώνα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκυγιόμ Μπαλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπουργέ, πριν από λίγες μέρες συζητούσα ε, με τη Γαλλίδα Υπουργό Εργασίας, την Υπουργό στην πατρίδα μου, και ρώτησα τι γίνεται σήμερα που αυξήθηκαν οι έλεγχοι στη Γαλλία, ε, τι γίνεται με την εσωτερική αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την απόσπαση των εργαζομένων και μου είπε ναι μεν αυξήθηκαν οι έλεγχοι, αλλά ακριβώ ε, λόγω αυτού βλέπουμε ότι είναι τεράστιο το έργο. Τώρα το καταλάβαμε δηλαδή που αυξήσαμε τους ελέγχους, δεν το είχαμε αντιληφθεί. Και εταιρείε που παραβαίνουν τον νόμο σήμερα είναι πολύ περισσότερες από εκείνες που υποπτευόμαστε. Και επέμεινε στο γεγονός και νομίζω ότι έχει δίκιο ότι υπάρχει έλλειψη ευρωπαϊκού συντονισμού για τον έλεγχο. Είναι απλό όμως βασικά και μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα. Και ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κανένα πρόγραμμα γι' αυτό θα κάνετε σημαντικές συνόδους ε, και συναντήσεις ε, κορυφής μεταξύ Υπουργών Εργασίας. Το έχετε στη μέση διάταξη, έχετε προτάσεις για καλύτερο συντονισμό των επιθερήσεων εργασίας και να πάμε να πιάσουμε τους παραβάτες, εκείνους που παραβαίνουν σήμερα τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Danke, jetzt Ευχαριστώ κύριε Ράιντκε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Εδώ κάθομαι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Επέστρεψα και εγώ από την Πρατισλάβα. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που μπορούμε να συζητάμε μαζί σας στα πλαίσια της Σλοβακικής Προεδρίας δύο ερωτήσεις. Η πρώτη μάλλον είναι μια έκκληση. Άκουσα και εσά και του συναδέλφου και βλέπουμε ότι η αναθεώρηση τη οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων δημιουργεί πολλέ ανησυχίε σε πολλού από εμά. Οποιαδήποτε και αν είναι η τοποθέτησή μα και ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτέ στην Επιτροπή μα, αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι ένα διαχωρισμό μεταξύ Ανατολή και Δύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το θέλουμε. Εργαζόμενοι λοιπόν στο Συμβούλιο αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια όχι μόνο αυτά τα οποία έχουν θέσει κίτρινη κάρτα, αλλά και τα κοινοβούλια εκείνα τα οποία δεν έχουν θέσει κίτρινη κάρτα, είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ε, συνεργασία που θα έχουμε, εσείς να καταφέρετε να συντονίσετε καλύτερα την όλη συζήτηση, προκειμένου να αποφευχθεί ο διαχωρισμός αυτός, η διχόνοια ή ο κατακαιρματισμός. Δεύτερη ερώτηση, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναφερθήκατε σε νέους από περιθεροποιημένες ομάδες. Το ζήτημα μας είχε απασχολήσει και εδώ, καθώς επίσης και σε συνεργασία που έχουμε με οργανώσεις νέων από όλη την Ευρώπη. Είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε στοχευμένες δράσεις για να αποφύγουμε περιθεροποίηση κοινωνικών ομάδων όπως η Ρωμά. Δεν ξέρω λοιπόν αν μπορούμε στα πλαίσια της αξιολόγησης πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και στα πλαίσια της αξιολόγησης της εγγύησης για τους νέους να ασχοληθούμε και με τις ομάδες αυτές όπως η Ρωμά. Έχει τελευταία μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Θα ήθελα να μάθω τις προθέσεις σας ως Προεδρία και πώς θα επιτύχετε συμβιβασμό για την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Είναι πολύ ακαθόδε το θέμα και πολύ σημαντικό για τη δική μου χώρα. Επίσης, τι γίνεται με την ε, νομοθεσία για την πρόσβαση, την προσβασιμότητα. Δεν έχει να κάνει μόνο με την επιβάρυνση οικονομική και διοικητική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό τι δουλειά έχει ε, η πρόσβασιμότητα και επιβάλληση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί αν μια επιχείρηση ή ένα κατάστημα είναι προσβάσιμο για όλους και για άτομα με αναπηρία, αυτό σημαίνει ότι θα έχει και περισσότερους πελάτες και περισσότερες δουλειές και περισσότερο τζίρο και περισσότερα κέρδη. Γιατί διαμαρτύρονται οι μικρομεσαίες ότι είναι ε, βάρος αυτό. Επίσης, και αυτή η ίδια η έννοια της προσβασιμότητας θα πρέπει να θεωρείται συνολικά. Δηλαδή αν υπάρχει στην αρχή ένα επιπλέον κόστος, αυτό όπως βαίνεται αρκετά ε, γρήγορα και εύκολα. Στις Ηνωμένε ε, Πολιτείες έχει αποδειχθεί ότι αυτό λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Και σας ερωτώ λοιπόν τι προθέσεις έχετε. Ακούω διάφορες δικαιολογίες για να μπλοκαριστεί αυτή η προσπάθεια. Τώρα αυτό είναι το καινούριο που ακούμε ότι είναι λέει κάτι που επιβαρύνει διοικητικά και οικονομικά τις μικρομεσαίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Βλέπετε, Υπουργέ, ότι εδώ στην Επιτροπή μας ασχολούμαστε με πάρα πολλά θέματα και ποικίλα. Και αν είχαμε και άλλο χρόνο θα μας ε, κατέβαιναν και άλλες ιδέες. Και τώρα έχετε παρακαλώ 22 λεπτά για να απαντήσετε όσο μπορείτε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι εξεπλάγει ευχάριστα ε, για το ότι η χώρα μου αναφέρθηκε πολύ συχνά και πολλοί δημοσιογράφοι μου είπαν ότι όταν έρθει στις Βρυξέλλες όλοι θα είναι διακοπές, όλα θα είναι άδεια, όμως ξεπλάγει. Υπάρχει πολλοί κόσμος εδώ που ενδιαφέρεται για τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε, που ενδιαφέρεται για τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Είναι λοιπόν ένα πολύ θετικό μήνυμα και είναι μια καλή αρχή για το πώ μπορούμε να αλλάξουμε την οτροπία ε, των Ευρωπαίων πολιτών και την αντίληψή τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τους στόχους της Προεδρίας μας είναι αυτός. Υπήρχαν πολλές ερωτήσεις, γι' αυτό λοιπόν ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων εάν δεν καταφέρω να απαντήσω στον καθένα από εσά ξεχωριστά. Θα προσπαθήσω να εστιάσω τι απαντήσει μου στι προτεραιότητες της Προεδρίας και να καλύψω έτσι τις ερωτήσεις σας. Εάν μετά έχετε και άλλες ερωτήσεις, με τα χαράς να μπω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσω λέγοντας ότι δύο χρόνια πριν αναλάβουμε την Προεδρία, είχαμε ήδη επικοινωνία με την τριπλή Προεδρία, κάτω χώρες, Σλοβακία και Μάλτα. Οι έξι μήνες είναι ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και είναι σχεδόν αδύνατον να αρχίσει κανείς να επεξεργάζεται ε, ένα θέμα και να το ολοκληρώσει. Για τον λόγο αυτό, και το τονίζω, το είπα άλλωστε και στην αρχή, θέλουμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Θέλουμε να ε, αναπτύξουμε τις ε, προτεραιότητές μας και να συνεχίσουμε αυτά που άρχισαν οι προηγούμενοι. Θέλουμε λοιπόν να δοθεί μια συνέχεια ε, στις προσπάθειες των ε, προηγούμενων προεδριών. Γι' αυτό λοιπόν ε, και μια που άκουσα ότι ο υπουργό της Μάλτας βρίσκεται εδώ, με τα χαρά να συνομιλήσω μαζί του για τα διάφορα θέματα που μας απασχολούν. Διότι σίγουρα δεν θα ολοκληρώσουμε όλα τα θέματα με τα οποία έχουμε καταπιαστεί σε αυτό το εξάμεινο. Αρχίζω λοιπόν με την ερώτηση που ετέθη για το πώς θα αλλάξουμε την αντιμετώπιση, την αντίληψη των Ευρωπαίων πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα γίνει αυτό. Θεωρώ προσωπικά και ταυτόχρονα αυτή είναι και η θέση της Προεδρίας της Σλοβακίας, ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να έρθουν πολύ πιο κοντά στους πολίτες. η νομοθετική και μη νομοθετική εξουσία είναι ε, κάπως αόρατη. Γι' αυτό λοιπόν και η Προεδρία μας θα διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις στη Σλοβακία, όπου οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί μας και εμείς να τους πουλήσουμε τα επιτεύγματά μας. Προσπαθούμε δηλαδή να εντείνουμε, να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες, διότι πιστεύουμε πως είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και να συζητηθούν εκτενέστερα, έτσι ώστε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τώρα, έλαβα πολύ καλά σχόλια για την άτυπη σύνοδο κορυφής, ιδιαίτερα για την ψηφιοποίηση που συζητήθηκε και τον αντίκτυπο αυτής στους ανθρώπους, στην αγορά εργασίας, στο εργατικό δίκαιο. Και μάλιστα το γεγονός και μόνο ότι το 90% των συμμετεχόντων ήταν υπουργοί, ήταν κυβερνητικοί, ε, μας δείχνει πόσο σημαντική είναι η ψηφιοποίηση και πόσο θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να βρούμε λύσεις στα μεγάλα ερωτήματα. Για παράδειγμα, προσωπικά μετά από 20 χρόνια στον πολιτικό στίβο, προσπάθησα μέσω άτυπων συνεδριάσεων, μέσω εκδηλώσεων να δράσω. Προσπαθήσαμε με επιτόπου επισκέψεις να δούμε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, να δούμε πώς έχει ε, αλλάξει η ρομποτική τη βιομηχανία, τι γίνεται στα εργοστάσια, πώς ε, και αν αντικατέστησαν τα ρομπό τους ανθρώπους, τι έγιναν οι απολυμμένοι. Ενδεχομένως τώρα μία διαφορετική αντιμετώπιση θα είναι κάτι που θα καλωσορίζαμε. Έχουμε θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους, γι' αυτό πιστεύω πως είναι σημαντικό να, να μην μείνουμε στα λόγια και να συνδέσουμε την θεωρία με την πράξη. Πήγαμε σε ένα εργοστάσιο στη Σλοβακία και είδαμε πώς αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αυτήν την μετάβαση. Και πιστεύω πως αυτή ήταν η σωστή προσέγγιση. Και νομίζω τώρα απαντώ εν μέρει και στις ερωτήσεις που μου κάνατε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση, πώς θα επιτύχουμε τους ε, στόχους μας, πώς θα έρθουμε πιο κοντά στους πολίτες. Αυτό πιστεύω πως δεν ισχύει μόνο για την Προεδρία μας, αλλά για όλα τα θεσμικά όργανα και νομίζω πως συμφωνούμε όλοι. βλέπουμε πως ο κοινωνικός διάλογος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε κοινωνικό, κοινωτικό επίπεδο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε συμβιβαστικό πνεύμα και αυτό μπορούμε να το δούμε και στην οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Είναι ένα θέμα που αφορά ε, για διαφορετικούς λόγους όλους μας. Γι' αυτό θα διοργανώσω ένα συνέδριο στην Πρατισλάβα για το θέμα αυτό. Σίγουρα δεν βλέπουν όλοι οι εργοδότες την οδηγία από την ίδια οπτική γωνία. Ακούμε για παράδειγμα ε, εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων στη Γερμανία που μας λένε ότι δεν έχει καμία απολύτως ε, χρήση, κανένα απολύτως όφελος αυτή η οδηγία. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί διαφορετικές απόψεις οι οποίες πρέπει να συζητηθούν ανοιχτά. Και αυτή θα είναι μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας, ανεξάρτητα από το αν θα μπορέσουμε να της δώσουμε ένα αίσιο τέλος. Σίγουρα πρέπει να συζητηθεί. Φυσικά και θα θέλαμε η οδηγία αυτή να μπορεί να υλοποιηθεί μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Όμως πρώτα έπρεπε να περιμένουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από τις 11 κίτρινες κάρτες από τα κράτη-μέλη που αφορούσαν την επικουρικότητα. Αυτό τώρα βρίσκεται υπό συζήτηση. Τώρα μπορεί να συνεχίσει η ομάδα εργασίας και να προχωρήσει στην έγκριση των μέτρων μετά, όπως σας είπα, σχεδιάζουμε διάφορα συνέδρια. Και ας μην ξεχνάμε και τις ε, χώρες Βίσεγκραντ, όπου συνεδριάσαμε και βρήκαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να βρούμε κάποιο κοινό τόπο. Τον Ιούνιο όταν έγινε μια σημαντική τροποποίηση, πιστεύουμε πως καλύτερο θα ήταν να περιμέναμε κάποιο χρονικό διάστημα από έξι έως 9 μήνες μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή, γιατί στο διάστημα αυτό ενδεχομένως να άλλαζαν γνώμη κάποια κράτη-μέλη. Όμως τώρα ό,τι έγινε, έγινε, έχει ληφθεί μια απόφαση, δυστυχώς χωρίς να ξέρουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στην πράξη. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ μέχρι τώρα στην Ευρώπη. Δηλαδή τα παλιά κρατημέλη απέναντι στα νέα Υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές θέσεις που βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι. Χρειάζεται λοιπόν ανοιχτός διάλογος, ανοιχτή ε, διάβλη επικοινωνίας και να ακούμε την άποψη των χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Να δούμε αν υπάρχει κάποια ευκαιρία για συμβιβασμό έτσι ώστε να εγκριθεί η οδηγία. Δεν αμφέβαλα ποτέ ότι είναι αναγκαία η οδηγία. Όμως πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε επί του περιεχομένου, έστω και συμβιβαστικά. Όταν συζητήσαμε τα θέματα αυτά, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά, με τον κύριο Γιούγκερ και την κυρία Τάισεν, στην πρώτη συνεδρίαση που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κυβέρνηση, το πρώτο που μου είπαν και η κυρία Τάισεν και ο κύριος Γιούγκερ ήταν το θέμα αυτό της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων. Και να μπω και σε κάποια πιο επίκαιρα θέματα επτά συγκεκριμένα, απαντώντας στις ερωτήσεις που κάνατε. Λοιπόν, ε, ε, νομοθεσία, πράξη για την προσβασιμότητα. Ποιο είναι εδώ το βασικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η Προεδρία μας. Είναι να έχουμε γενική πρόσβαση του κοινού παντού. Αυτό θα προωθήσουμε στο Συμβούλιο. Η ουσία της πρότασης είναι πάρα πολύ περίπλοκη και χρειάζεται πάρα πολλές διαβουλεύσεις και τακτικές προσπάθειες συντονισμού και στα ίδια τα κράτη-μέλη. Η Προεδρία μας φιλοδοξεί να συνεργαστεί και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να διαδραματίσετε εσείς ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Και χαίρομαι πολύ που βλέπω ενδιαφέρον και ανταπόκριση από πλευρά σας. Ελπίζω στο μέλλον αυτό να φανεί και από συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ίδιο ισχύει και με τα άλλα θέματα. Έρχομαι στα υπόλοιπα ζητήματα που θέσετε. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο συμπεριλαμβάνει πολλά συγκεκριμένα πράγματα σε κάποιους τομείς της οικονομίας Ακούσαμε και για το Brexit. Εγώ περιμένω πολλά από τη Σύνοδο Κορυφής ε, των Ευρωπαίων Ηγετάων στην Πρατισλάβα. Ξέρω ότι ο Πρωθυπουργό μας είναι σε επαφή και με άλλους ηγέτες και είναι αισιόδοξο. Και για την υποστήριξη ε, των νέων και την καταπολέμηση της ανεργίας τους που είναι και αυτή μια πολύ μεγάλη πρόκληση που θα συζητήσει και αυτή η Σύνοδος Κορυφής. Δεν θα αναλωθεί στο Brexit. Θέλουμε να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τους πολίτες μας και τους νέους μας και ίσως με κάποια μέτρα θετικής διάκρισης έτσι ώστε να βρίσκουν δουλειά. Έρχομαι τώρα στην απόσπαση εργαζομένων ξανά. Σας είπα, πολλά θέματα έχουν σχέση με αυτό. Έχω προσωπικές διαβουλεύσεις ε, κατηδίαν με τους συναδέλφους μου υπουργού. Εγώ είμαι φύση αισιόδοξο και νομίζω ότι το Δεκέμβριο ε, δεν είμαι ακόμα σε θέση να σας πω ότι θα έχουμε μια καλή οδηγία και θα έχουμε καταλήξει. Αυτό θα ήταν μάλλον Ε, Θα πρέπει να συνεχθούμε και με τους κοινωνικούς εταίρους που έχουν εδώ πολύ σπουδαίο ρόλο να παίξουν. Εμείς στη Σλοβακία, βέβαια έχουμε την εθνική μας θέση και την υπερασπιζόμαστε, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας για να μεσολαβήσουμε και να φέρουμε σε αίσιο πέρα την όλη υπόθεση, δηλαδή να εγκριθεί η οδηγία. Για τον κοινωνικό πυλώνα και τα κοινωνικά δικαιώματα στα οποία αναφερθήκατε, περιμένω εδώ να εγκριθεί μια κοινή προσέγγιση και να υιοθετηθεί για την κοινωνική προστασία, για τα κοινωνικά δικαιώματα και τα εργασιακά. Από σας είπα, εισαγωγικά, υπάρχει και κάτι ακόμα η ατζέντα, το θεματολόγιο για τις νέες δεξιότητες. Θα πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή, γιατί αλλάζει ραγδαία η αγορά εργασίας. Μεγαλύτερη ψηφιοποίηση, διαβίου, μάθηση κτλ. Δεν μπορούμε εμείς να επαναπαυόμαστε. Αρκεί να ανατρέξουμε στην ιστορία και να θυμηθούμε ε, το κίνημα ε, ε, των λουδιστών, λουδιτών, συγγνώμη, οι οποίοι κατέστρεφαν τις μηχανές, γιατί θεωρούσαν ότι όταν εμφανίστηκαν οι μηχανές στα εργοστάσια θα τους έπαιναν τις δουλειές. Τώρα δεν μπορούμε εμείς να βγούμε να καταστρέφουμε τα ρομπότ. Λόγω της ψηφιοποίησης ε, θα υπάρχει κόσμος που θα απολυθεί, αλλά θα πρέπει να μετακπαιδευτεί σε κάτι ε, νέο για να μπορεί να βρει δουλειά σε ένα νέο περιβάλλον ε, ψηφιοποιημένο και να συνάδει με τις νέες ε, τεχνολογίες. Θα υπάρξουν συστάσεις λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή κατά τη διάρκεια της προθέσης μας. Στην Πρατισλάβα ήδη συζητήθηκε αυτό το θέμα. Ενδεχομένω 400 εκατομμύρια άνθρωποι ε, θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν λόγω της ψηφιοποίησης και της απώλειας των θέσεων εργασίας τους. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, άλλο θέμα, και ο συντονισμός τους. Σας είπα και εγώ προηγουμένως, καθυστερήσαμε γιατί περιμέναμε το δημοψήφισμα. Αν είχε βγει άλλο αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα ξέρουμε πώς εξελίχθηκε το δημοψήφισμα και θα πρέπει οι ηγέτες να δώσουν μια ευθεία απάντηση για το τι σχέση θέλουμε να έχουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται ένας συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλες οι ε, αλλαγές θα πρέπει να λαμβάνονται ε, υπόψη. Εργασία και απασχόληση των νέων. Και σε αυτό αναφέρθηκα ήδη εν μέρη. Έχει σημασία για μας αυτή τη στιγμή να συνεχίσουμε να ε, βοηθούμε τους νέους να προσπαθούμε να βρούμε και άλλους πόρους για την υποστήριξη. Υπάρχουν κάποια κονδύλια. Υπάρχουν κονδύλια για την αντιμετώπιση ενεργείας των νέων. Πριν από δυόμιση χρόνια η ανεργία των νέων ήταν πολύ μικρότερη στη χώρα μου, σήμερα έχει φτάσει στο 24%. και τα κονδύλια έχουν μειωθεί. Αλλά δεν έχει σημασία τόσο πολύ να δούμε πόσα χρήματα αφιερώνονται εκεί, αλλά αν πιάνουν τόπο. 84% των νέων που βρήκαν δουλειά μέσω των κονδυλίων αυτών διατηρούν τη δουλειά αυτή. Δηλαδή, 84% των νέων, επαναλαμβάνω, διατήρησαν τη δουλειά τους και από την εκπνοή των προγραμμάτων και μετά. Είναι σημαντικό λοιπόν γιατί βοηθούν τους νέους να βρουν μια δουλειά και μετά ακόμα και όταν διακόπτονται ή εκπνέουν υπάρχει ε, μόνιμη θέση αποσχόλησης για τους νέους. Δεν μπορώ να εξαντλήσω όλα τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε, ούτε να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν απάντησα επαρκώς. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, με χαρά να το κάνω. Με, πολλές από τις προτάσεις είναι νομοθετικές Ορισμένες θα συζητηθούν στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου, Συμβούλιο Υπουργών ε, Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας και θα αρχίσει η διαδικασία υλοποίησης κάποιων νομοθετικών ε, προτάσεων. Αυτά είναι θέματα ειδικών, θα συζητηθούν στην Βρατισλάβα και εγώ θέλω να ενημερώνονται οι πολίτες όσο γίνεται περισσότερο για να καταλαβαίνουν ε, τι ρόλο ε, διαδραματίζουν τα διάφορα θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκτενή σας απάντηση. Νομίζω ήταν καλή συζήτηση. Ελπίζω να μην είναι η τελευταία που θα έχουμε μαζί σας κατά τη διάρκεια της Σλοβακική Προεδρίας. Τώρα σε λίγο θα ψηφίσουμε για τη θέση μας για τον προϋπολογισμό του 2017. Αναφερθήκατε σε αυτό. Έχουμε ένα σχέδιο του Συμβουλίου με μεγάλες περικοπές σημαντικές, ιδιαίτερα σε εκείνες τις θέσεις και τα κονδύλια που μας ενδιαφέρουν εμάς, δηλαδή καταπολέμηση ενεργείας των νέων, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καταπολέμηση της φτώχειας κτλ. Στην πρωινή συζήτηση για τον προπολογισμό Όλα τα μέλη της Επιτροπής που μίλησαν ε, εκφράστηκαν σαφέστατα προς την εξής κατεύθυνση. Επειδή είναι προτεραιότητες όλα αυτά τα πράγματα και επίγουσες, χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Τώρα θα αποφασίσουμε τη δική μας θέση και θα σας παρακαλούσα να μας υποστηρίξετε στο Συμβούλιο είναι σημαντικά αυτά τα κοινωνικά ζητήματα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας παρακαλούμε να φροντίσετε να πάρουμε περισσότερα κονδύλια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε και άλλες γενιές να πάνε χαμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε τη δική σας υποστήριξη και θα σας είμαστε ευγνώμονες αν το προωθούσατε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. So, Μικρό διάλειμμα.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 So, können wir dann... Λοιπόν, μπορούμε να αρχίσουμε με τις πληροφορίε. So, ich rufe auf den Tagesordnung. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 11 της ημερησίας διάταξης. Γενικός προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, όλα τα τμήματα. Έχουμε το κατάλογο της ψηφοφορίας όλοι και μπορούμε να αρχίσουμε. Συμβιβαστική τροπολογία D. 5677. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε 5678. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνατε. 5602. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 5602. έξι μηδέν όλοι. μία ψήφος παραπάνω για το ΕΛΚ και για την ECR. Παρακαλώ, ρυθμίστε. Εντάξει, τώρα βγάλαμε τη μία. Ψηφίσατε. Όχι. Απορρίπτεται. Μαριαν Χάρκιν. Ναι, ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη και από τα μέλη της Επιτροπής. Ξέχασα την κάρτα ψηφοφορίας. Λυπάμαι, ειλικρινά. Γι' αυτό λοιπόν ε, ας το λάβετε αυτό υπόψη στις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Καμιά φορά ξεχνιέται κανείς, το συγχωρούμε, αλλά μία φορά στον καθένα. Δεν αλλάζει βέβαια αυτό το αποτέλεσμα. Για την 5602 απορρίπτεται και πάλι. Περνάμε στην 5657. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5603. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 5603. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. 5604. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 5604. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 5637. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5605, υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε ηλεκτρονικά, 5605, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 56-22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56-38. Τα σχόλια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5606. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5607. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 5607 ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 56-40. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 56-40. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία Α5674. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56-59. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 56-09. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56-10. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 56-10. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. 56-39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56-11. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 56-11. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Β. 56-75 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά, αν και νομίζω είναι προφανές το αποτέλεσμα. Συμβιβαστική Β. Πέρας. Απορρίπτεται. 56-12 υπέρ. Κατά. Νομίζω πως απορρίπτεται. 56-60 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 56, 69 και 56, 28 τις έχουμε τακτοποιήσει. Περνάμε στην 56, 33. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 56, 13. Υπέρ. Ξανά 56-13. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56-14, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56-15, figures, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56-15, remarks με προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56-17. Υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεν βλέπω τα χέρια σας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Προφανώς εγκρίνεται. 56-62 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 56-62 remarks υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56-18 figures υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56-18 remarks, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56-68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία όχι, με συγχωρείτε, λέει ο προεδρο 56 56-19. Με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. Κατά, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική C. 56-76. Υπέρ. Κατά. Κατά, Εγκρίνεται. 56-42. Υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 56-21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56-23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56-73 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56-29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56-56. Όχι, καταπίπτει. 56-31 5631, λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56-32, με προφορική τροπολογία, figures, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56-32, remarks, με προφορική τροπολογία του εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 56-35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56-43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56-55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56-55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56-63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν πολλές τροπολογίες τώρα και τελειώσαμε. Τελική ψηφοφορία δεν νομίζω πως χρειάζεται, διότι είναι προφανές. Τελειώσαμε λοιπόν αυτή τη ψηφοφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ακολουθεί η επόμενη λογικά. Έχουμε και κατάλογο ψηφοφορίας εδώ στο σημείο 12. Λοιπόν, βλέπετε όλο αυτό το μακροσκελή τίτλο. Εφαρμογή της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Γενικής Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά στις 21 Μαΐου 2012 όπως τροποποιήθηκε στι 8 Μαΐου 2013 ε, για την εφαρμογή της Σύμβασης τη διεθνού οργάνωση εργασία του ΕΠΤΑ σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλληλείας. Το ξέρω ότι τώρα έχω επισύρει τη μήνυ των διερμηνέων που δεν με προλάβανε. Ε, τώρα, 7 σειρέ τίτλο, επικεφαλίδα έκθεση, καιρό έχω να δω για να είμαι ειλικρινή. Καταλάβατε όλοι τι πράγμα πρόκειται και τι θα ψηφίσουμε. Το 12 είναι, βάση περιπτώσει, παράγραφος 1, τροπολογία 12 είπε. Κατά. Απόχες. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, ας αλέξουμε. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Για να δούμε τι έχουμε. Απορρίπτεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική ε. Πάμε στην τροπολογία 16 υπέρ κατά νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Αμφιβάλλει κανεί Όχι. 19 υπέρ. Κατά. Αυτό θέλει έλεγχο. Η 19 παρακαλώ γιατί δεν είναι σαφές. Δεν σηκώνεται χέρια ή δεν τα βλέπω εγώ. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 26-26 ισοψηφία. το λοιπόν. Ανθρωπολογία 20. Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η συμβαστική β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική σ υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε την τροπολογία 7 υπέρ. Όχι, είναι μέσα στη συμβαστική. Δεν εγκρίθηκε η δι. Τελειώσαμε τότε. Εγώ φταίω, λέω πρόεδρος, έκανα λάθος. Πάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Σας παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Μάλιστα. Πέρες ψηφοφορίας. 46 υπέρ. 6 κατά, χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγητρία. Das Ergebnis kommt an den Bericht. Διαφωνεί κανείς με την έκθεση, ε, όχι. Ο Τόμας Μαν. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστήσατε τον εισηγητή της τελευταίας έκθεσης, αλλά νομίζω θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τον προηγούμενο εισηγητή, έναν Τόμας Χέντελ εδώ για τον προπολογισμό. Εξαιρετική έκθεση. Λοιπόν, επόμενο θέμα στην ημερησία δέξη παριθμό 13. Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη. Η συγητής είναι ο Όλε Κρίστενσεν. Πριν του δώσουμε το λόγο, παρακαλώ οι διμερείς επαφές και συζητήσεις και τα πηγαδάκια να διεξαχθούν εκτός της αιθούσης στο λόμπι εδώ απ' έξω. Bericht sollte schon noch jemand da bleiben. Καλά, ας μείνει και κανένας για την έκθεση, δεν <laughs> είπαμε να διάσει η αίθουσα. So, λοιπόν, στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη. Θα μας ενημερώσει για όλα αυτά ο κύριος Όλε Κρίστινσεν και έχει αμέσως το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που δίνετε το λόγο. Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σχετικά με τη στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη. Είχαμε ένα στενό διάλογο με διάφορους συμμετέχοντες στον τομέα των αερομεταφορών. Ήρθα σε επαφή με ανθρώπους που συμμετέχουν στον κλάδο αυτό, στις δικαλιστικές οργανώσεις, στο κατασκευαστικό κλάδο και συζητήσαμε με τους ενδιαφερόμενους πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε δίκαιες συνθήκες εργασίας στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές και πρόωθησα βέβαια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις παρατηρήσεις τους. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνένεση ανάμεσα στους διαφερόμενους. Θεωρούν ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές για να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τον κλάδο αυτό και για να διατηρήσουμε θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη. Ω συντάκτη γνωμοδότηση είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια επικοδομητική γνωμοδότηση με συγκεκριμένε δράσει, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα δίκαιο μέλλον για του ανθρώπου που ασχολούνται στον τομέα αυτό. Ασχολούμε με πέντε σημεία τα οποία θα πρέπει να μα απασχολήσουν προκειμένου να πετύχουμε το δίκαιο αυτό μέλλον στο οποίο αναφέρομαι. Κοινωνικό διάλογος καταρχά Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν ισχυροί ανεξάρτητοι κοινωνικοί εταίροι στο τομέα τη αεροπορία. Πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία διαβούλευση και ενημέρωση να ενισχυθεί ο κοινωνικό διάλογο στο συγκεκριμένο κλάδο. Η μείωση στην συμμετοχή συνδικαστικέ οργανώσει αποτελεί πλήγμα κατά του κοινωνικού διαλόγου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υφίσταται το δικαίωμα για τη συγκρότηση και τη συμμετοχή στη συνδικαλιστική οργάνωση, ότι αυτό είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο απασχόλησε είναι τα νέα μοντέλα απασχόληση τα οποία προέκυψαν την τελευταία δεκαετία. Μολονότι ορισμένα χρησιμοποιήθηκαν για μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερο ανταγωνισμό, αλλά έχουν οδηγήσει περισσότερο σε μια αναζήτηση ευνοϊκότερη νομοθεσία από ορισμένα κράτη-μέλη ή από ορισμένε επιχειρήσει. Καταλαβαίνετε ότι η δινή αυτή χρήση ορισμένων νομοθεσιών βάλει κατά τον ανταγωνισμό, αλλά ακόμα και τι ίδιε τι ασφάλεια και των προτύπων ασφάλεια. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να απαγορεύσουμε τις συμβάσεις μηδενικών ορών εργασίας καθώς επίσης και τα καθεστώτα pay to fly. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να αποσαφενιστεί το κριτήριο έδρα βάσης. Έπειτα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι συμφωνίες υπάρχουν με τρίτες χώρες και στα πλαίσια των συμφωνιών αυτών θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Αναφέρομαι τέλος στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης Τομέα πάρα πολύ σημαντικό για όλη την αλυσίδα προστιθέμενη αξία των αερομεταφορών. Επίση είναι πολύ σημαντικό να γίνονται οι απαραίτητη χρηματοδότηση των προγραμμάτων έρευνα και εκπαίδευση. Τέλο, αναφέρομαι και στο ζήτημα τη υγεία και τη ασφάλεια. Όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυτό θα πρέπει να έχουν σε ασφαλείς συνθήκε εργασία ανεξάρτητα από το μέγεθο τη εταιρεία που του απασχολεί. Ανεξάρτητα από το πού εργάζονται και τι είδου σύμβαση έχουν. Υποστηρίζω λοιπόν το ότι θα πρέπει όλες οι αεροπορικές εταιρείες να υπάγονται σε συγκεκριμένες επιθεωρήσεις όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Δεν μπόρεσα να κάνω και άλλες τροπολογίες, επειδή όπως ξέρετε πρέπει να συμμορφωθούμε με συγκεκριμένο αριθμό λέξεων όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις μας. Προσβλέπω πάντως τις θετικές και επικοδομητικές παρεμβάσεις των υπόλοιπων συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Όλε. Συζήτηση από το ΕΛΚ, ο κύριος Κόχ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή Όλε Κρίστενσεν. Πολύ καλή γνωμοδότησή του ήδη. Καλό είναι, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν συγκρούσεις αρμοδιοτήτων ε, μεταξύ ΕΜΠΛ και ΤΡΑΝ, για την έκθεση για το κοινωνικό dumping. Ε, ευχαριστώ που κατάφερε να επικεντρωθεί στα κοινωνικά ζητήματα. Ε, αναγνώρισε και διαπραγματεύτηκε, τα, διαπραγματεύτηκε μάλλον τα ε, σημαντικότερα ζητήματα και είμαι βέβαιος ότι από κοινού μπορούμε να συνεχθούμε και να βελτιώσουμε τη γνωμοδότηση. Από την αρχή της δεκαετίας του 90 που απελευθερώθηκαν οι αερομεταφορές έχουν γίνει πολλά. Ε, αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ε, ιδιαίτερα αν δούμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες ε, είναι εκτεθειμένε σε παγκόσμιο ανταγωνισμό που δεν γίνεται σε καμία περίπτωση με τρόπο θεμητό πάντα. Με τη νέα στρατηγική Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θέλει να αντιμετωπίσει τη διεθνή κατάσταση και να ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων με ποιοτικέ μεταφορές και προδιαγραφέ και πρότυπα για του επιβάτε. Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση και να έχουμε ποιοτικές θέσεις εργασίας και στις αεροπενταφορές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε νέα μοντέλα επιχειρησιακά, επιχειρηματικά, όπως το pay to fly που πληρώνει ε, ο εργαζόμενος για να ε, είναι υπτάμενος και το σημείο 4 τα αναφέρει αυτά και νέα μοντέλα απασχόλησης τα οποία δεν είναι όμως πάντα αρνητικά. Δεν θα πρέπει να τα απαγορεύσουμε καταρχήν και από χέρι, αλλά να τα ρυθμίσουμε και να προβλέπουμε συγκεκριμένα μέτρα ε, που να εγκυώνται μεγάλες ε, προδιαγραφές και ψηλά πρότυπο. Χαίρομαι που στο σημείο 5 της γνωμοδότησης κάνει λόγο εισηγητής για την ιδιαίτερη ε, κατάσταση των υπερβολικά κινητικών ε, εργαζομένων και θα πρέπει να υπάρχει κάποια βάση ε, που είναι η έδρα των εργαζομένων αυτών ε, και η πατρίδα τους. Είμαστε ακόμα σε μια μεταβατική περίοδο δεκαετή που δεν είναι υποχρεωμένες οι εταιρείε να εφαρμόζουν αυτή την ιδέα της βάσης και της έδρας του εργαζομένου και προτείνω λοιπόν να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και τακτική ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κράτων μελών και κοινωνικών εταίρων. Έτσι ώστε να αναγνωρίζουμε νωρίς νέες ε, τάσεις απασχόλησης εργοδότησης και να φροντίσουμε να επικρατούν σωστές συνθήκες. Γενικά, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη μετακπαίδευση και στην διαβίου εκπαίδευση και παρακατάρτιση. Ε, το σημείο 8 δεν το προσέχει πολύ αυτό. Θα πρέπει να έχουμε εργαζομένους έμπειρους, ε, ε, καλά καταρτισμένους και γι' αυτό ζητώ να είναι πανεπιστημιακού επίπεδου εκπαίδευση, ε, με διτή εκπαίδευση στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν και νέα δεδομένα με νέα αεροσκάφη όπως είναι τα drones, τα μη επανδρομένα και ε, άλλες ε, εξελίξεις τεχνολογικές. Θα κάνω σχετικά τροπολογία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Σλοτκόφσκι από το e ΙΣΙΑ. Άλτε, δεν έχω συγγετή και πάλι. Έχω. Έχω. Τα πάμε και το πρωί αυτά. Ε, είναι δεύτερη φορά που μου πέφτει ο κλήρος, αλλά εγώ είμαι τώρα. Τι να κάνουμε. Καταρχάς, ε, ευχαριστούμε πολύ τον για την έκθεση και πιστεύω πως θα αποτελέσει πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση. Στα πλαίσια της νέας στρατηγικής για την Ευρώπη, η ασφάλεια, ειδικά στον χώρο των μεταφορών και των αερομεταφορών, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να δοθεί λοιπόν βάση στην ασφάλεια, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην μετεκπαίδευση. Δυστυχώς έχουμε εύλογους λόγους να πιστεύουμε ότι ορισμένες πρακτικές των αεροπορικών εταιρεών έχουν ε, δυσμενείς επιπτώσεις. Καταρχάς, χρησιμοποιείται το pay to fly πρόγραμμα, όπου οι πιλότοι δηλαδή πρέπει οι ίδιοι να πληρώνουν τις ώρες πτήσης και την εκπαίδευσή τους. Και οι πιλότοι ως, ε, ως αποτέλεσμα εργάζονται περισσότερες ώρες για να μπορέσουν να τα επεξέλθουν οικονομικά. Και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρηματολόγησε όταν ε, ζητήσαμε πληροφορίες πως ε, δεν έχει λάβει ε, λεπτομέρειες σχετικά με, την, με τον αντίκτυπο της πρακτικής αυτής. Αυτού του τύπου η απασχόληση είναι ευρέως διαδεδομένη στις, στην αεροπορία και Σύμφωνα με μία μελέτη, το πρόγραμμα Pay to Fly θα πρέπει να απαγορευτεί όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παγκόσμια. Χρειάζεται μία νέα στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη, έτσι ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ειρήνα Ρωνιακάρη για την Κούρε έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτήν την πολύ καλή έκθεση. Πιστεύω ότι συμφωνούμε. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία χρειάζονται επίλυση και υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την επίλυση αυτή. Δεν είμαι απόλυτα πεπισμένη για την ε, ορθότητα της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα αποφύγουμε το κοινωνικό dumping στις αερομεταφορές. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση εκεί και μάλιστα στην Επιτροπή μας είχαμε και επισκέπτες, πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους οι οποίοι ε, εκπροσωπούσαν τον κλάδο και μας είπαν πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν. Πολλές φορές οι πιλότοι αναγκάζονται να δουλέψουν άρρωστοι γιατί κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους εάν δεν εργαστούν. Αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες ε, συνθήκες. Πτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να εξετάσουμε μεγάλη προσοχή ε, το τι συμβαίνει, όπως και τις, ε, τις συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν θα επιμείνω ότι η αφετηρία μας θα πρέπει να είναι οι αεροπορικές εταιρείες, οι ευθύνη που έχουν εκείνες. Μόνο υπό συγκεκριμένε προϋποθέσεις θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή αλλού. Χρειάζεται επίσης ε, να ορίσουμε τι σημαίνει ακριβώς η έδρα βάσης, το home base. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των εργαζόμενων. Χρειάζεται πραγματικά να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όμως ε, θα ήθελα να παρακαλέσω να δώσουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να μπορέσουν τα ίδια να καταπολεμήσουν τα ε, προβλήματα. Πολλές φορές ε, βλέπουμε πως αεροπορικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε χώρες όπου δεν έχουν ακόμα λάβει άδεια ε, εργασίας. Είναι πολλά τα προβλήματα. Τα pay to fly πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και είμαι σίγουρη ότι μετά από τη συζήτηση στην Επιτροπή θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Λάουρα έχει το λόγο, η οποία όμως λείπει. Η Ζωέλ Μελάν τότε. Ζητώ συγγνώμη. Ε, την Καριμάντελή ε, δεν ε, βλέπω που έπρεπε να λάβει το λόγο. Η Τζιν Λάμπερτ θα αναλάβει εξ ονόματο των Πρασίνων. Ναι. Την αντικαθιστώ την κυρία Ντελή που είναι σκιώδη μα για αυτό το θέμα. Και εκείνοι, όπως και άλλοι, θα ήθελα να ευχαριστήσουν τον εισηγητή για την πλήρη γνωμοδότησή του που καλύπτει τα βασικά σημεία του θέματος και πάλι το θέμα των επισφαλών θέσεων εργασίας είναι σημαντικό για μας και μεγάλη απειλή για την ασφάλεια ενεργητική και παθητική στην αεροπορία. Την τελευταία δεκαετία βλέπουμε τους ψευδοαπασχολούμενους, ε, συμβόλαια μηδενικών ωρών, συμβόλαια που πληρώνει ο κυβερνήτης για να πετάει είναι κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Βλέπουμε νέες μορφές επισφαλών θέσεων εργασίας. Θα πρέπει αυτές να εξαφανιστούν για να είναι όσο δυνατό υψηλότερο το επίπεδο ασφαλείας για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες. Υπάρχει αυτό το στοιχείο το ανθρώπινο ε, στις επισφαλείς μορφές εργασίας και θέσεις σε ε, τομείς πολύ ευαίσθητους ε, όπως είναι οι αερομεταφορέ και θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί οι αεροπορικέ τραγωδίες όπω η πρόσφατη τη German Wings. Ε, θα συνεργαστούμε, χαιρόμαστε που ο εισηγητή ζητεί να τερματιστούν οι ε, συμβάσεις που αναφέρονται στο σημείο 4 και βεβαίω η άμεση απασχόληση, η κανονική απασχόληση θα πρέπει να είναι ο κανόνα για να αποφεύγονται και το κοινωνικό dumping. Προσβλέπουμε συνεργασία με τον συντάκτη τη γνωμοδότησης έτσι ώστε οι εφαίρες μας να είναι ασφαλείς και για τους εργαζομένους στις αεροπορικές εταιρείες αλλά και για τους επιβάτες. Και το θέμα της έδρας ε, και της βάσης ε, θα θυμάστε τις προσπάθειες που είχαν γίνει από μια συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία όταν αναθεωρήσαμε το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν θα την αναφέρω γιατί ε, ε, μας έχουν πει να μην μιλάμε για αυτούς εδώ μέσα στην Επιτροπή μας ε, και έχει βάλει έδρα για πολλούς εργαζομένους μια χώρα που ήταν πολύ χαμηλές οι εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν ζούσαν καν σε αυτή τη χώρα. Άρα όλα αυτά τα θέματα είναι ε, ε, γνωστά, θα πρέπει να τα δούμε όμως εγκάρσια σε όλα τα νομοθετήματα για να υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια ε, στα όσα λέμε. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η Τζιν εννοούσε τη Ryanair φαντάζομαι, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος ότι είναι αυτή η εταιρεία. Η κυρία Τζέα κανονικά θα είχε τώρα το λόγο, αλλά δεν τη βλέπω στην αίθουσα. Η ευθυντή Ουδής Τώρα η κυρία Μελά από την ΕΝΕΦ. Όχι, δεν ζήτησα το λόγο, λέει η κυρία Μελά. Δεν κατάλαβα. Δεν θέλετε να μιλήσετε. Όχι, όχι. Ζητώ συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι λέγατε. Όχι, δεν θα μιλήσω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Ωραία. Η Μαρίτα Ούλφσκοκ τότε. Yes. Uh, thank you first of all. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ τον συντάκτη της γνωμοδότησης, τον Όλε, για την γνωμοδότηση αυτή που επικεντρώνεται στα βασικότερα σημεία που θα πρέπει να απασχολήσουν την Επιτροπή μας, την Επιτροπή Απασχόλησης. Υπάρχουν βέβαια ορισμένα σημεία τα οποία θα ήθελα να τονίσω λίγο περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα για τον κλάδο των αερομεταφορών και κυρίως για την κοινωνική πτυχή της ε, στρατηγικής για τις αερομεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πτυχή αυτή είναι ακόμα πολύ αδύναμη. Χαίρομαι που βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί με το κοινωνικό διάλογο. Πρέπει να υποστηριχθεί ο κοινωνικό διάλογο στον κλάδο των αερομεταφορών. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πιλότοι αλλά και πληρώματα εδάφου και αέρου που δεν είναι καν σε θέση να οργανωθούν συνδικαλιστικά και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν συμβάσεις που δεν επιτρέπουν στους εργαζόμενους να ενταχθούν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτό είναι απαράδεκτο και προφανώς παραβιάζει τις συμβάσεις ε, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Χρειαζόμαστε όμως μεγαλύτερη δέσμευση και περισσότερες δράσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου πραγματικά να έχουμε καλές συνθήκες απασχόλησης σε αυτόν τον κλάδο. Αυτό που θα μπορούσε επίσης να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει τις ε, συνθήκες απασχόλησης είναι να ενισχύσει το ευρωπαϊκό, μάλλον την Ιάσα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, η ΆΣΑ, θα πρέπει να έχει περισσότερους πόρους και μια ευρύτερη εντολή, προκειμένου να μπορεί να ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά. Θα πρέπει να γίνει μια τροποποίηση προφανώ του καονισμού τη. Δεν πρέπει να μιλάμε για ασφάλεια αν δεν υπάρχει επαρκή επίβλεψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε πάρα πολλά συμβάντα χωρίς όμως να υπάρχουν καθόλου υπάρχει ανάληψη δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ορισμένε περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε δράση όταν έβλεπε ότι υπήρχε παραβίαση τη νομοθεσία, αλλά ακόμα και αυτό δεν αρκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει επίση ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, στα πλαίσια του οποίου μπορούν να δραστηριοποιούνται οι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Και ακούσαμε και το παράδειγμα μια μόνο εταιρεία, υπάρχουν και πολλέ άλλε που δεν ακολουθούν τους κανόνες του θεμητού ανταγωνισμού. Πέρα από όλα αυτά και ολοκληρώνοντας πρέπει να σας πω ότι η άμεση απασχόληση θα πρέπει να παραμείνει η συνήθις μορφή απασχόλησης στις αερομεταφορές. Πρέπει να επιμείνουμε στο σημείο αυτό και θα πρέπει να διευρύνουμε αυτή τη στιγμή την απέτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει μόνο με ένα 50% θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό των άμεσα απασχολούμενων και να έχει να κάνει όχι μόνο με τους πιλότους αλλά και με το προσωπικό εδάφος και αέρους. Ξέρετε ότι δώσαμε μάχες πραγματικά με την Ryanair αλλά και με άλλες αεροπορικές εταιρείες και υπάρχει τουλάχιστον μία εταιρεία που μετά την παρέμβαση της ΕΑΣΑ δεν μπόρεσε να συνεχίσει τις δραστηριότητές της και χρειάστηκε να συμμορφωθεί. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην επιτρέψουμε, ειδικά για τον κλάδο αυτό, να διέπεται τελικά από πρακτικές αθέμητες, όπου δεν θα υπάρχει καμία απολύτως ρύθμιση για λόγους ασφάλειας αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμόζεται κοινοτική νομοθεσία και θα μπορούσαμε μέσω της νομοδότησης του ΟΛΕ να θέσουμε πραγματικά αυτές μας προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ζος Μπάχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους ε, συναδέλφους που ευχαρίστησαν και συνέχαραν τον ε, Όλε για την πολύ καλή έκθεση. Ο κύριος Κρίστενσεν μας ανέφερε πως είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και εγώ το βρίσκω ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι πολύ φιλόδοξη η έκθεση και Νομίζω πως κατάφερε να, ε, τουλάχιστον στην αφετηρία να το καταφέρει. Υπάρχουν βέβαια κάποιες προκλήσεις όσον αφορά το πόσο φιλόδοξη θέλουμε να είναι αυτή η στρατηγική. Εδώ θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δείξει την ε, προσοχή που θα έπρεπε, δεν ήταν όσο τολμηρή έπρεπε ο κοινωνικός διάλογος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, κομμάτι της έκθεσης και τον χαιρετίζω. Ιδιαίτερα ο διάλογος με τις τρίτες χώρες και τις ε, προδιαγραφές και τους κανονισμούς της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας. Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντική αναφορά ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό. Σίγουρα θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την έκθεση σε λεπτομέρειες. Είναι άλλωστε το πρώτο σχέδιο αυτής. Το σημείο 3 μου αρέσει πάρα πολύ που αναφέρεται στην ασφάλεια και στις ε, ασφαλείς συνθήκες απασχόλησης. Οι συνάδελφοι επίσης αναφέρθηκαν στο σύστημα Pay to Fly, στην ε, έδρα της ε, αεροπορικής εταιρείας, στη σημαία φέρει εταιρεία. Είναι όλα πολύ σημαντικά όσον αφορά το κοινωνικό ντάμπινγκ. Πρέπει επίσης να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή και να ζητήσουμε συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με την έδρα βάσης. Και τέλος θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον όλες. Το σημείο 6 μας αναφέρει ε, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, ξένους εργαζόμενους. Τι ακριβώς εννοεί. Ε, σε γενικέ γραμμέ, πιστεύω πως είναι πολύ καλή η έκθεση και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους για τις καλές παρεμβάσει τους. Πιστεύω πως είμαστε πολύ φιλόδοξοι και αυτό φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κριστόφ Τριζάρ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση MOVE, έχει τώρα τον λόγο. Thank you, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο να πω Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Επιτροπή σα ε, επιλαμβάνεται αυτού του θέματος, πάρα πολύ σημαντικό για τη στρατηγική για τις αερομεταφορέ. και βλέπουμε από τι πρώτε συζητήσει ε, ότι συμφωνείτε κι εσείς με τις προτεραιότητες και τα ε, βασικά ζητήματα για μας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για ό,τι επιθυμείτε και προσβλέπουμε στη μελλοντική συνεργασία μας για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όλε εσύ έχεις τον τελευταίο λόγο. Όχι γενικώ για την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ ε, για όλα τα σχόλια. Πραγματικά ε, πολύ καλά ε, παντρεύονται με αυτά που έλεγα και εγώ στην γνωμοδότησή μου. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους που το ανέφεραν ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην έχει προχωρήσει αρκετά και συμφωνώ και εγώ και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι που θα καλωσορίζαμε και καλωσορίζουμε. Αλλά Τώρα έχουμε την ευκαιρία να αντιδράσουμε αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνική στρατηγική και για τις αερομεταφορές. Γιατί μέχρι τώρα ε, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, διαπιστωνόταν έλλειμμα σίγουρα θα βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε πολύ καλές προτάσεις ε, σε ό,τι μας αφορά ως Επιτροπή απασχόλησης. Συμφωνώ πάρα πολύ ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση για να έχουμε ε, πεπειραμένους και ε, καλά εκπαιδευμένους εργαζομένους που μας χρειάζεται ακριβώς για να ενισχυθεί η ασφάλεια των αερομεταφορών θα δώσω ίσως μεγαλύτερη προσοχή. Και σε σχέση με την έδρα και τη βάση, αυτό θα πρέπει να ισχύει πραγματικά, διότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες όταν μετεκαθίστανται σε τρίτες χώρες, χρησιμοποιούν εργαζομένους εκεί, αλλά σήμερα δεν χρειάζεται καν να μετεγκατασταθούν και το λέω αυτά στο Ζορς παραμένουν στην Ευρώπη και εκεί μπορούν να απασχολούν ε, εργαζομένους από τρίτες χώρες ως ευρωπαϊκό εργοτικό δυναμικό, διότι έχουν έρθει εδώ πλέον αυτοί. Υπάρχουν άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή ε, και ε, είναι σε αθέμητο ανταγωνισμό με τις δικές μας. Θα πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να εξασφαλίσουμε ένα θεμητό και δίκαιο ανταγωνισμό και ίσους ε, όρους του παιχνιδιού. Ευτυχώς έχουμε πολλές εταιρείες αξιόλογες που κάνουν πολύ καλή δουλειά, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μερικές που προσπαθούν να παρακάμπτουν τους κανόνες, να τους διαστρεβλώνουν, να τους ε, φέρνουν στα μέτρα τους. Κανείς δεν το είπε εδώ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω εκείνους που ισχυρίζονται ότι δίνουμε δουλειά στον κόσμο. Το γεγονός ότι δίνεται δουλειά σε πολύ κόσμο δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι έχει κανείς και τη σωστή συμπεριφορά επειδή απασχολεί πολλούς εργαζομένους. Χρειάζονται λοιπόν οι κανόνες παιχνιδιού για όλες τις εταιρείες. Βεβαίω μπορεί να είσαι ανταγωνιστικό στην τιμή, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπουλάμε και τα πάντα. Χρειάζεται ε, δίκαιος ε, και θεμητό ανταγωνισμό παντού. Έτσι λοιπόν, χαίρομαι για τη μελλοντική μας συνεργασία και είμαι ε, βέβαιος ότι θα καταλήξουμε με τη βοήθειά σας σε μια πολύ καλή έκθεση. Σας ευχαριστώ για όλα τα επικοδομητικά σας σχόλια. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Νομίζω ότι τελειώσαμε το σημερινό μας πρόγραμμα. Το 14 είπαμε ε, σημείο αναβάλλεται για λόγους ε, χρονοδιαγράμματος άλλης επιτροπής. Άρα σήμερα σχολάμε λίγο νωρίτερα. Ε, καλή σας μέρα, απόγευμα και βράδυ και θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9. Χαίρετε.